Good morning everybody who will start. Καλημέρα σε όλες και όλους. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα τα πω ισπανικά από εδώ και πέρα. El primer punto del orden del día es adopción de, de la agenda. Eh, si estamos... Καταρχάς, σημείο 1 έγκριση σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Ε, να σας πω ότι το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης ε, θα το συζητήσουμε μετά από το σημείο 8. Έχετε αντίρρηση κατά τα λοιπά. Όχι, εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών. Έχετε στο φάκελό σας ε, τα πρακτικά. Φαντάζομαι ότι τα έχετε διαβάσει. Υπάρχουν προβλήματα. Ναι, κυρία Μπέλτριχα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει δερμηνία στα αγγλικά. Vamos a Τώρα, ε, εντάξει. Bueno, Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά τα οποία ε, ψνάπτονται στην μέση διάταξη. Περνάμε στο επόμενο σημείο ανακοινώσει τη Προέδρου. Όπως γνωρίζετε, στις 25 Νοεμβρίου είναι η διεθνή ημέρα κατά της βίας ε, λόγω φύλου. Και θα συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία από τα Ηνωμένα Έθνη για τις γυναίκες ε, μούντο ναράχα, κόσμος πορτοκαλί ε, για τις ε, γυναίκες. Ε, θα φωτιστεί λοιπόν πορτοκαλί και το κοινοβούλιο. Έτσι θα συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερη ανακοίνωση, να σας πω ότι στις 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο με ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Θέμα οι προτεραιότητες ε, της ισότητας των φύλων ε, στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερσιάς διάταξης που είναι η ώρα ψηφοφορίας. Έχετε φαντάζομαι μαζί σας τις κάρτες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Καταρχάς ψηφίζουμε την ε, γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2014. Η κυρία η συγκέντρια θέλει το λόγο, συντάκτρια μάλλον. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως όλες και όλους τους συναδέλφους, μέλη της Επιτροπής ε, των Γυναικών και για την υποστήριξή τους αλλά και για όλες τις ε, τροπολογίες άριθμες ε, που έχουν καταθέσει για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα για το οποίο η Επιτροπή μας συντάσσει γνωμοδότηση και για την ΤΕΒΕ είχαμε και η Ντρουά που είναι η επίσης αρμοδιεπιτροπή συνέταξε. Τώρα Αφού ευχαριστήσω όλους, θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες και τους συμβούλους και να πω ότι υπήρξε ένα γεγονός σημαντικό που το ξεπεράσαμε μένα, αλλά ελπίζω να μην αποτελέσει συνήθι πρακτική εκ μέρους ελιστικής ομάδας. Δηλαδή την τελευταία στιγμή, την ενδεκάτη ώρα να πω, αλλάζουν κάποιους συμβιβασμούς και περιπλέκουν ιδιαίτερα τα πράγματα. Ευτυχώς ε, καταφέραμε με μια προφορική τροπολογία να σώσουμε την κατάσταση. Σας παρακαλώ ε, ταπεινά σε οποιαδήποτε άλλη ε, παρόμοια περίσταση να με ενημερώσετε εκ των προτέρων και όχι την τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ την κυρία Μπεθερλή και μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 42. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία την οποία υπέβαλε η κυρία Ροντρίγκε υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Πρώτο κομμάτι όμως, σε δύο τμήματα. Πρώτο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία για το δεύτερο κομμάτι. Θα ε, το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε τις τροπολογίες 50. Ψηφίσαμε. Μήπως θα πρέπει να ξανακάνουμε την ψηφοφορία, την επαναλαμβάνουμε για το δεύτερο τμήμα, να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα κιόλα. Πέρα της ψηφοφορίας. De acuerdo. Hay... Ωραία. 14 ψήφους κατά γιατί ένας βουλευτής των Πρασίνων που δεν έχει την κάρτα μαζί του καταψήφισε την πρόταση. Τέλο πάντων, το συμπέρασμα είναι ότι απορρίπτεται το δεύτερο κομμάτι. Πάμε στην τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52, δύο τμήματα, δύο τμήματα. Το πρώτο κομμάτι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει μια τροπολογία προφορική, η 53, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Sí, la enmienda 54 también hay que votarla. ¿Votos a favor? Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 61 σε δύο τμήματα, το πρώτο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 61 υπέρ εγκρίνεται 15 υπέρ 12 κατά και μία αποχές τροπολογία 63 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ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 εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 σε δύο τμήματα. Πρώτο κομμάτι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 σε δύο τμήμα, πρώτο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψηφίσατε. Απορρίπτεται η τροπολογία. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 σε δύο τμήματα, στο πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 σε τρία τμήματα αυτή τη φορά. Πρώτο κομμάτι, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 σε δύο τμήματα ή όχι. Α, όχι, καταπίπτει. Όχι δεν θα ψηφίσουμε την 68 ούτως ή άλλως διότι υιοθετήθηκε η τροπολογία 97. Εξού και περνάμε στην 98 ε, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται, 99 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμών 1. Κυρία Αρένα, μήπως θα μπορούσα να ζητήσω ένα διάλειμμα για την ομάδα μου για δύο δευτερόλεπτα. Α, μας λείπει μια σελίδα στον ε, κατάλογο των ψηφοριών. Θα a dar dos minutos. Αντί δύο λεπτά διάλειμμα. Vale, eh, Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Βρισκόμαστε στην τροπολογία υπαριθμών 1. Την ελέγξαμε? Όχι, τώρα. Θα ψηφίσουμε... λοιπόν, ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Είπαμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 1 πάντα. Cierra la votación. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά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 Το ελέγχουμε την 16 ηλεκτρονικά. Πέρα τη Απορρίπτεται η 16. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο κομμάτι υπέρ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 ε, καταπίπτει η προφορική τροπολογία 2. Τώρα περνάμε στην προφορική τροπολογία 1 σε δύο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. Δεύτερο κομμάτι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την ε, γνωμοδότηση. Ε, ξεκινάμε. Πέρας της Εγκρίνεται με 23 ψήφους ε, υπέρ, 6 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, Στην κυρία Μπέκερη Λιμπάριο. Y pasamos a la siguiente votación. Eh. στη δεύτερη ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότηση τάση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία ΤΙΣΑ. Συμβιβαστική υπαρθμόν 3, ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική υπαρθμόν 4, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31. Έχουμε μια προφορική τροπολογία από την κυρία Νόχελ. Έχει ληφθεί υπόψη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν καταλαβαίνω. Καλό είναι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να βεβαιωθούμε για το αποτέλεσμα. Τροπολογία 32 πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 34. Απροβάδα. Εμείνα. εγκρίνεται. Σημαστική 5 υπέρ. Μάλλον 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα η συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Σε la Πέρας ψηφοφορίας. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, Α, έχει αποσυρθεί. Withdraw. Τώρα συμβαστική 7. εν Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε 55. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 14 ήταν οι αντίθετε ψήφοι. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 59 ψηφίσατε όλοι απορρίπτεται. Τροπολογία 60 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Είναι αμφίροπο το αποτέλεσμα. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της 61 παρακαλώ. εγκρίνεται 15 υπέρ 14 κατά. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 62, όχι δεν θα ψηφιστεί γιατί είναι γλωσσική φύσεως. Πάμε στην 63 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ θέλετε να ελέγξουμε να ελέγξουμε την 70 άρχεται η ψυχοφορία. πέρας Δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Πολύ γρήγορα μπόρεσα και μέτρησα. Όχι, τυχαίο ήταν. Δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Λοιπόν, ε, συμβαστική ένα υπέρ κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ως προσθήκη με προφορική τροπολογία από την κυρία Νόιχελ ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι δεν θα το διακινδυνεύσω να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Τροπολογία 3. Έγκριντ. Τροπολογία 5 με προφορική τροπολογία από την κυρία Ζητνάνσκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 10 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω εκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε τροπολογία 12, έρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπεβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το σύνολο ως έχει αποποιηθεί. Άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση 20 ψήφι πέρα 9 κατά καμιά αποχή. ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Έχουμε ολοκληρώσει σήμερα τις ψηφοφορίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε και η συνεδρίασή μας. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Con respecto al informe de opinión de Έχουμε την εφαρμογή και επανεξέταση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Ασίας. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκέρλιν. Να περιμένουμε όμως δύο λεπτάκια. Bueno, pues vamos a Να ah, συνεχίσουμε λοιπόν τις ε, εργασίες της Επιτροπής μας, παρακαλώ. Αν υπάρχει κάποιο πηγαδάκι, παρακαλώ εκτός εθούσης, γιατί εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Το επόμενο λοιπόν σημείο στην εμείς διάταξη, όπως είπα, είναι η εφαρμογή και επανεξέταση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Ασίας. Με εισηγήτρια η συντάκτρια γνωμοδότηση σε συγκεκριμένη περίπτωση, την κυρία Τζούλη Γκέρλιν. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο για να μας παρουσιάσει τις ιδέες της. Παρακαλώ κύριε Γκέρλιν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη γραμματεία για τη βοήθεια που μου παρήχαν ώστε να συντάξω αυτή τη γνωμοδότηση. Επίσης και τους σκιώδεις, δεν έχουμε συναντηθεί βέβαια ακόμη, αλλά περιμένω να συνεργαστούμε όμορφα. Όσοι από εσά δεν γνωρίζετε καλά την Κεντρική Ασία, έχει πέντε ανεξάρτητες χώρες, Καζακστάν, Τατζικιστάν κτλ. Η Κεντρική Ασία είναι γεωγραφικός χώρος, ε, ρίζες έχει στην περσική κουλτούρα και γλώσσα και είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό ιστορικά διότι ε, αυτό χαρακτηρίζει και τις συμπεριφορές. Πρόκειται για γνωμοδότηση προς την ΑΦΕΤ που συντάσσει σχετική έκθεση για τη στρατηγική της ε, στην Κεντρική Ασία. Δεν μπόρεσα βέβαια να βάλω όσα θα ήθελα σε αυτή τη γνωμοδότηση καλωσορίζω οποιαδήποτε τροπολογία. Δηλαδή σίγουρα χρειαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά επειδή η Κεντρική Ασία συναποτελείται από πέντε ανεξάρτητα κράτη ε, με τις δικές τους κουλτούρες, είναι δύσκολο βέβαια να ε, συλλογικά εκπροσωπήσουμε τις επιτυχίες και τα προβλήματα. Η βία εναντίον των γυναικών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αν και έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ, 29% των γυναικών στην περιοχή είναι θύματα σεξουαλικής βίας πρέπει να παροτρύνουμε τις διοπτικές αρχές να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με αυτό το θέμα και θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες για να ενισχύσω αυτό το σημείο. Ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν μεγάλες ανησυχίες για τη βία κατά των γυναικών και η εμπορία των γυναικών είναι ανησυχητική. Έχουμε αυξητική τάση σε δύο κράτη. Υπάρχει ένας ρόλος εδώ που θα μπορούσε να παίξει ο συντονιστής και να βοηθήσει περισσότερο γιατί αν θέλετε έχουμε μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι βάλωτος είτε επειδή είναι φτωχός είτε επειδή είναι εκτεθειμένος άμεσα στην οικιακή βία. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτών των κρατών. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω τις διοκτικές αρχές αυτές της χώρες να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προ... πολλές προκλήσεις και προβλήματα στην περιοχή, αλλά θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένα θετικά. Έχει υπάρξει πρόοδος. Δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε, αλλά βεβαίως η πρόοδος αυτή δεν επαρκεί. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δεχτούμε ότι έχει υπάρξει. 58% αυτών που αποσχολούνται στο γεωργικό τομέα στην Κεντρική Ασία είναι γυναίκες. Οι γυναίκες παίζουν κρίσιμο ρόλο στη γεωργία. Λοιπόν, θα με ενδιέφερε να ξέρω τι ποσοστό αυτών των γυναικών γεωργών είναι ιδιοκτήτες της γης. Θα υποβάλω λοιπόν σε σχέση με τη γεωργική ιδιοκτησία και τον ρόλο των γυναικών ε, τροπολογίες. Ακόμη Υπάρχει και ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που θα ήθελα να υπογραμμίσουμε. Μέχρι πρόσφατα οι άντρες του Κύρκισταν θα μπορούσαν να απαγάγουν την ε, γυναίκα που θέλουν να παντρευτούν. Ε, δεν ήταν έγκλημα, ήταν παράδοση αυτό. Εμείς τώρα ε, έχουμε συνηθίσει κάποιος να μας ζητά το χέρι γονατιστός. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό από το να αρπάζεις τη γυναίκα που θέλεις δεν πρόκειται για έγκλημα καθόλου στο Κυρκυστάν. Πέρσι βέβαια τροποποίησαν τον νόμο, το σχετικό και έγινε αδίκημα ποινικό η απαγωγή της ε, νύφης που θέλουν. Βεβαίω οι νόμοι μεταβάλλουν την συμπεριφορά αλλά δεν την μεταβάλλουν μέσα σε μια νύχτα. Συνεπώς υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, η τροποποίηση του δικαίου είναι σωστό βήμα, βέβαια, αλλά αν ασχοληθούμε στη γνωμοδότησή μας με αυτό το θέμα θα έπρεπε να υποστηρίξουμε αυτούς στο Κυργιστάν που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου ώστε να γίνει πραγματική συμπεριφορά. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια από τους σκιώδεις και για να συνεργαστώ ε, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα θέλατε. Eh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκέρλιν για την παρουσίαση. Και τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Γκίρλινγκ για αυτή τη θαυμάσια γνωμοδότηση. Δίνει πολλέ πληροφορίε, έχει θετική προσέγγιση, παροτρύνει προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι σωστή αυτή η τοποθέτηση προς τρίτες χώρες. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες που διατυπώνονται ως προς τη βία κατά των γυναικών. Πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα των δικαίων, του των δικαιωμάτων ενώπιον του δικαίου και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα οι γυναίκες να συμμετέχουν στην οικονομική πρόοδο. Θα προσέθεσα τέσσερα στοιχεία την συμμετοχή των κοινωνικών στο δημόσιο βίο ε, και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, η καταπολέμηση των στερεοτύπων από πολύ μικρή ηλικία, τρίτον, η εφαρμογή των στρατηγικών που ήδη υφίστανται και τέλος, θα ήθελα να επιμείνω ότι είναι αναγκαίο για μας να συνεχίσουμε να έχουμε έναν διάλογο και ακόμη και αν έχουμε στοιχεία τα οποία είναι ανησυχητικά, αναφέρομαι στο σημείο του κειμένου που λέει ότι ανησυχούμε ότι μία γυναίκα στις τρεις είναι θύμα βίας, θα ήθελα να σας μεθυμίσω ότι στην Ευρώπη έχουμε την ίδια αναλογία περίπου. Συνεπώς εδώ δεν δίνουμε μαθήματα, απλώς θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος και να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για να αποδώσουν καρπούς. Είναι τα τέσσερα στοιχεία λοιπόν που κατά την άποψή μου είναι σημαντικά και θα ήθελα να τα προσθέσω αυτά τα στοιχεία με τη μορφή τροπολογιών. Θα ήθελα όμως να συγχαρώ την κυρία Γκέρλινγκ για αυτή τη γνωμοδότηση που είναι πλούσια σε περιεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκάμπριελ εκ μέρους τώρα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η κυρία Αρενά έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω κι εγώ στην αξιολόγηση της εκθέσης κυρίας Κλούλη. Είμαστε στην Επιτροπή των Γυναικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να με τα ζητήματα της νομιμότητας κατά τρόπο σαφή όσον αφορά τις ε, χώρες Κεντρικής ε, Ασίας, διαβάζοντας τις εκθέσεις των ΕΕ και της ε, ΟΑΣΕ βλέπουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις, πρέπει να τις σημειώσουμε, τις θετικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται. Προτείνω 11 τροπολογίες, 4 τυπολογικές σκέψεις και τροπολογίες στο διατακτικό ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των συμβάσεων των Εθνών για την απάλληψη κάθε μορφή διακρίσεων ει βάρο των γυναικών. Ζητούμε από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να αναπτύξει ένα σχέδιο δράση για την ισότητα των φύλων. Ζητούμε να αναπτύξουν τα κράτη τη Κεντρική Ασία αποτελεσματικέ πολιτικέ για να αποτρέψουν κάθε τύπο διακρίσεων ει βάρο των γυναικών. Εν γέννη δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα στην κατεύθυνση που ζητούμε πάντα κατά των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Ευχαριστώ. Άλντε τώρα. Κυρία Μπέρντερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω και εγώ και θα ευχαριστήσω την κυρία Γκέρλιν για τη δουλειά της. Είναι πάντα δύσκολο όταν ε, συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες, χώρες με διαφορετικές ε, παραδόσεις και νοοτροπίες. Να είμαστε επιθετικοί εμένα, αλλά όχι ε, να υποδεικνύουμε επιλογές. Δεν πρέπει δηλαδή να ξεπερνούμε τα εσκεμένα και τις, ε, τους όρους της ε, αυροφροσύνης ε, στην ανθρώπινη συμπεριφορά. ξέρετε ότι σε ορισμένε κοινότητε μπορεί κάποιε τι υποδείξει να έχουν αποτελεσματικότητα, αλλά όχι πάντα. Και πρέπει πάνω απ' όλα να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική προστασία των γυναικών. Εκεί ε, ιδιαίτερα το ζήτημα των νυφών που παραγγέλλονται διαλληλογραφίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διάχυση τέτοιων ζητημάτων σε όλο και πιο απομαξιμένες περιοχές της υπαίθρου και πρέπει να εξασφαλίσουμε το, ίδιο, το είδος εκείνο της προστασίας το οποίο θα μπορέσει να καταρρύψει ε, παραδοσιακές αντιλήψεις εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση, υπάρχουν δυνατότητες για διαζύγιο και ούτω καθεξής. Και βέβαια και σε αυτό έχει επίσης εμπλακεί ιδιαίτερα και ασχοληθεί το Κοινοβούλιο, είναι η καταναγκαστική εργασία γυναίκες, παιδιά σε ε, βακοπαραγωγή, αναγκαστική και σε βέβαια ε, καταστάσεις όπου ξέρουμε ότι είναι αναγκασμένες να το κάνουν γιατί οι άντρες τους, οι πατεράδες τους έχουν φύγει στο Πακιστάν για να μαζέψουν τον μπαμπάκι στο Πακιστάν και εκείνες μένουν στην πατρίδα τους. Αυτά όλα πρέπει να τα κοιτάξουμε λοιπόν στις επαφές μας με τις τρίτες χώρες, να προβάλλουμε και τις αξίες μας και να κοιτάζουμε την νομική διάσταση πάντα. Καλές λοιπόν οι τροπολογίες και νομίζω ότι μπορούμε όλες μαζί να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Al respecto de... Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις για την έκθεση αυτή, δεν ξέρω αν η κυρία Γκέρλιν θέλει να δευτερολογήσει αφού άκουσε τις συντρόφισσες από τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος συμφωνών να συμπεριληφθεί η διαδικασία λήψη τελικών αποφάσεων, <coughs> δημόσια ζωή. Και βέβαια τα ζητήματα τα σχετικά με την απάλληψη των διακρίσεων είναι σχετικά, θα τα συζητήσουμε, θα βρούμε λύσει. Αυτό που θα ήθελα πράγματι να κάνω κατά την κατάρτιση αυτής της γνωμοδότησης θα ήταν να ε, εντοπίσουμε δύο-τρία πολύ σημαντικά θέματα στα οποία όλοι συμφωνούμε πάνω στα κύρια θέματα για να μπορέσουμε και να εξασφαλίσουμε την υιοθέτησή τους μέσα από την έκθεση της ΑΦΕΤ. Όχι όμως μακροσκελής καταλόγους. Δεν θα ήθελα δηλαδή μια λύση τύπου χριστουγεννιάτικου δέντρου που ο καθένας έβαζε ότι του αρέσει μέσα. Αυτό που ακούω από τη σκιώδη συζήτηση σήμερα νομίζω ότι με καθυσυχάζει και επιβεβαιώνει θα μπορούσαμε να βρούμε λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρλινγκ. Όπως είπαμε και στην αρχή της συνεδρίασης, έχει αλλάξει μερικές διάταξη. Οπότε μετά το 8 έχουμε το υπαριθμόν 11 σημείο που αφορά την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη, την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Η συγγήτρια μάλλον είναι η κυρία Μάλιν Μπιέρκ. Τη δίναμε στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Είναι όντως ε, πολύ σημαντική η ακρόαση που έχουμε προβλέψει για την ε, σώματεμπορία, για την κίνηση ανθρώπων. Έχουμε να κάνουμε με συνθήκες διαβίωσης έχουμε να κάνουμε με διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Δύο τροπολογίες, ιδιαίτερα φέρω να αναφέρω, οι περισσότερες είναι καλύτερες γιατί εμβαθύνουν περισσότερο, ενσωματώνουν τις διεθνείς συμφωνίες ε, και στο θεματολόγιο των ΗΠΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις συμφωνίες κατά της σωματεμπορίας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τις ε, προτάσεις τροπολογιών και να τις προσκαλέσω στις 19 Νοεμβρίου από τις 2 ε, έως τις 3 σε μια συνεδρία συντονιστών, ε, σκιωδών μάλλον, για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Αλλά θα ήθελα να ακούσω πρώτα τις σκιώδεις παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιέρκ. Είμαστε στο ΕΛΚ, η κυρία Λεγκρίπ. Oui, merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εν συντομία, αυτή τη στιγμή θέλω να υπενθυμίσω δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι εμείς σαν ΕΛΚ θα θέλαμε η γνωμοδότηση αυτή να μην αποτελέσει ε, ένα, μια, ένα έμνασμα για να αμφισβητήσουμε τις εμπορικές ε, πρακτικές. Ε, θα μπορούσε ενδεχόμενα να φανεί κάποια στιγμή ότι το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο αποτελεί την πηγή όλων των κακών. Ενώ εμείς στο ΕΛΚΑ πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια λογική εμπορική πολιτική και δυναμική εμπορική πολιτική η οποία θα μπορέσει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας. Δεύτερο στοιχείο, υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή Γυναικών ε, δεν ε, είχε, βέβαια δεν είχα, το είχαμε συζητήσει σε μια προηγούμενη γνωμότητα του 2010, το έχουμε πει, αλλά τέλος πάντων εμείς σαν Επιτροπή Γενικών δεν έχουμε στη διάθεσή μας σαφείς μελέτες και συγκεκριμένες με αριθμητικά στοιχεία για τις συνέπειες ε, της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής στην κατάσταση των γυναικών. Αυτό ήταν μία από τις τροπολογίες που είχα υποβάλει, δηλαδή να προσπαθήσουμε να έχουμε συμπληρωματικές αξιολογήσεις και μελέτες για το θέμα. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες για το ίδιο θέμα και χαίρομαι γι' αυτό. Υιοθετήσαμε βέβαια μια θέση, μια στάση ανοιχτή ε, επικοδομητικής συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της, ε, ε, των διαπραγματεύσεων για, την, για, τον ε, συμβιβασ... για, τον, για την διαμόρφωση ενός συμβιβασμού, μια συμβιβαστικής πρότασης και εμείς σαν ΕΛΚ θα θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συμβαστική πρόταση όμως θέλουμε σαν ΕΛΚ να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, ε, όχι ρεαλιστική, όχι ουτοπική, ε, ρεαλιστική πρόταση. Ευχαριστώ. Με ανθρωπιστική διάσταση πάντα. Ευχαριστούμε κύριε Λεγκρίπ. κυρία Γιάλα Σέντερ τώρα έχει το λόγο του μέρους ομάδας Σοσιαλιστών των Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από αυτά που άκουσα έμεινα λίγο αμήχανη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπιόρκ για την ε, πρόταση. Είναι μια καλή αφετηρία το κείμενό της και νομίζω ότι με τροπολογίες μπορούμε να ενισχύσουμε ορισμένε ε, πτυχές. Η κυρία Σαΐφη στην πρώτη της έκθεση μπορεί να μην είχε συμπεριλάβει κάποιες πτυχές γιατί είχε ε, γνώμη της Επιτροπής αλλά επειδή τη γνωρίζω και έχουμε συνεργαστεί, για θέματα που άπτονται της ισότητας. Νομίζω είμαστε στο μήκο κύματο, στο ίδιο πνεύμα. Κάτι είπε η κυρία Λεγκρίπ, ε, και τα μέσα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το έχουν ε, αναλύσει τι επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών που δεν ε, είναι ισορροπημένες ή δεν έχουν αυτά τα, ε, τις διατάξεις για υποχρεωτική εφαρμογή της ρήτας των δικαιωμάτων. Αλλά είναι ένας βασικός πυλώνας, όπως και η προστασία του περιβάλλοντος. Eh, Έχουμε σε λίγε εβδομάδε και την COP21 για το κλίμα στο Παρίσι, άρα προσλαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα με αυτή την έκθεση ε, μπορούμε να ε, ανακτήσουμε την ευκαιρία που χάσαμε το 2010 και έτσι να ζητήσουμε ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Διότι ναι, μεν οι εμπορικέ συμφωνίε δεν είναι διάβολο με κέρατα, αλλά δεν είναι και αυτές καθεαυτές, αν δεν έχουν αυτές τις υποχρεωτικές ρήτρε, ε, δεν είναι, παραλαμβάνω, και συμφωνίες που μπορούν να προωθήσουν ε, τομείς ε, που οι γυναίκες εκεί είναι οι περισσότερες εργαζόμενες, μεταπίτικη βιομηχανία, γεωργικές εργασίες, δικαιώματα ε, χρήση της γης, εκπαίδευση κτλ. κτλ. Και έχουμε και την εγκάρσια ρήτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε υποβάλει εμείς ορισμένες τροπολογίε ω ομάδα με στόχο πρώτον πάντα στο πνεύμα της κυρία ΑΕΦΗ του 2010. Δηλαδή να δοθεί υπαχρεωτικό χαρακτήρα στις ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις περιβαλλοντικές ρήτρε που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών που να προστατεύουν τις ευρωπαϊκές αξίες, αυτές οι ρήτρε και να τις προωθούν μέσα των εμπορικών συμφωνιών. Δηλαδή να αξιοποιούμε τις εμπορικές αυτές συμφωνίες ε, όχι μόνο για την οικονομική όθηση και ανάπτυξη αλλά και για την ε, ανθρώπινη ανέλυξη. Έχουμε λοιπόν καταθέσει τροπολογίες με τις οποίες ζητούμε υποχρεωτική ε, συμπερίληψη των ρητρών ανθρώπινων δικαιωμάτων, παραλαμβάνω και περιβαλλοντικών ρητρών που έχει ε, επικυρώσει και εγκρίνει η Ένωση. Έχουμε και τι σχετικέ ε, διατάξει του Διεθνού Σχολείου Εργασία κτλ. Να συμπεριλαμβάνονται λοιπόν οι ρήτρε στι εμπορικέ συμφωνίε, καθώ και ρήτρε σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία τη γη, την υγεία. Και αυτέ και αυτοί τομεί επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις ε, εμπορικέ συμφωνίες είναι ευάλωτοι οι γυναίκες ε, και μαζί με αυτές και οι οικογένειές τους. Επίσης είναι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας εφαρμογής δηλαδή αυτής της εγκάρσης ρήτρας κάτι που επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη για να εξασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτή η ρήτρα θα επηρεάσει τις εμπορικές συμφωνίες που ε, διαπραγματεύεται η Ένωση με τρίτες χώρες. Επίσης, για να πετύχουμε αυτό τον υποχρεωτικό χαρακτήρα θα πρέπει να γίνει και μια ανάλυση εκ των προτέρων και εκ των υστέρων για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν οι συμφωνίες αυτές ε, στις γυναίκες, ε, στις αυτόχθονες κοινότητες που ξέρουμε ότι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι γυναίκες. Θα πρέπει να γίνει αυτή η μελέτη πιστεύω. Νομίζω ότι συμφωνώ σε αυτό που είπε η κυρία Λεγκρίπ από αυτού, γιατί ναι, δεν υπάρχουν μελέτε, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν συστηματικά και υποχρεωτικά αυτή την ανάλυση, την εκ των και των υστέρων ανάλυση, να την ε, εφαρμόσουμε και στι ε, συμφωνίε τι εμπορικέ και να λαμβάνουμε υπόψη την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την περιβαλλοντική πτυχή. Και αυτό θα μα δώσει και τεχνογνωσία σημαντική στο κοινωτικό δίκαιο. Βέβαια χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση να βρούμε δείκτες αναφοράς για να μπορέσει να γίνει αυτή η μελέτη αντικτύπου σε αυτές τις εκ των προτέρων των υστέρων αναλύσεων των εμπορικών συμφωνιών και επίσης επαναλαμβάνω μια σημαντική ρήτρα είναι και η συμμετοχή των οργανώσεων των γυναικών ιδίως εκεί όπου ε, έχουν πετύχει ε, επιτεύγματα, έχουν ε, σημειώσει πρόοδο αυτές οι οργανώσεις των ε, γυναικών, μικροπιστώσει, χρηματοδότηση και η ΕΤΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνει υπόψη αυτέ τι χρηματοδοτήσεις για να βοηθήσει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επειδή επηρεάζει του διαπραγματευτέ, θέλω να εκφράσω τη λοιπόν που ακόμη και στο πιο πρόσφατο έγγραφο της Κομισιόν του Οκτωβρίου, δηλαδή 2015, για αυτά τα ζητήματα δεν ε, συμπεριλαμβάνεται ακόμη εγκάρσια ρήτρα. Άρα και ο υποχρεωτικό χαρακτήρας. Η υποχρέωση συμπερίληψη αυτών των μελετών. Θα πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο πολλή κυρώσεων. Ευχαριστώ. Αν δεν δηλαδή ε, υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται αυτέ οι ρήτρε. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει, υπάρχουν. Δεν βλέπω, με συγχωρείτε. Κυρία Φορέντσα. Eh, eh, Ήθελα να ευχαριστήσω την Μαλίν Μπιόρκ, την ε, συντάκτρια της νομοδότησης ε, και όλους όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Εγώ είμαι υπεύθυνη για την έκθεση στην Ίντα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Γυναικών, διότι αυτή η κατεύθυνση προς την οποία δουλεύουμε δείχνει ότι όσον αφορά την ισότητα των φύλων, όλο το θέμα αυτό δηλαδή της, ε, των ρητρών της, ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για έναν λόγο, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για να ζητήσουμε εκθέσεις ε, και μελέτες ε, αξιολόγησης εξπόστο και εξάντε, δηλαδή να εντάξουμε αυτή την ε, προοπτική την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και γι' αυτό ευχαριστώ την Επιτροπή Γυναικών και συμφωνώ ότι όντως θα πρέπει να ζητήσουμε, πρέπει να απαιτήσουμε μελέτες και θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να προωθήσουμε τα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση την, με την εμπορική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Muchas gracias, señora Εάν δεν υπάρχουν ε, άλλε παρεμβάσει, ε, δεν ξέρω αν η κυρία Μπιόρκ ε, θέλει να πάρει το λόγο για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους τους, όλες τις κοιότητες συζήτριες. Θα διατυπώσω τις προτάσεις, τις συμβαστικές. Είναι πολύ καλές προτάσεις σας και θα τις ενσωματώσω. Και ελπίζω ότι έτσι θα κερδίσουμε και την υποστήριξη του εισηγητή. Θα τα πούμε και στους συνεδρίες των σκιωδών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ζητήσατε το λόγο, αλλά θέλω να είστε πάρα πολύ συντομή γιατί θα έχουμε και την ακρόαση που ξεκινάει. Η Κομισιόν, η Κομισιόν θέλει να μιλήσει συγκεκριμένα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα είμαι σύντομη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή σα για τη σκληρή δουλειά που έκανε πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι το σχέδιο γνωμοδότησης όπω και σε άλλες περιπτώσεις καλύπτει όλε τι απόψει κληθεί όσον αφορά το θέμα της διάστασης των φύλων ενισχύει τους σωστούς μηχανισμούς, προωθεί την ενσωμάτωση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει τους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορούμε, η Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω αυτά τα θέματα ε, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που υφίστανται όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στοιχείων, τις επιπτώσεις των συμφωνιών των εμπορικών, τι εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών και τι θα έπρεπε να ε, περάσει στο θέμα της συνεργασίας. Ε, έχουν υποβληθεί ε, τροπολογίες, μια προσπάθεια να αποσαφηνίσουν αυτό το θέμα. Ορισμένες τροπολογίες μοιάζουν να μην λαμβάνουν υπόψη τους πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική και θα ήθελα να σας πω ότι η Κομισιόν είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσει με οποιαδήποτε συνεισφορά σε σχέση με αυτό το θέμα. Muchas gracias, pues, eh, finalizado. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, ξεκινάμε την ε, ακρόαση, όμως κάνουμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα ένα μισή-δύο λεπτά, έτσι ώστε ε, όλοι όσοι πρέπει να μπουν στην αίθουσα να πάρουν τις θέσεις τους και μετά θα ξεκινήσουμε.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 Eh, λοιπόν, ξεκινάμε αυτή την ακρόαση για την ε, διάσταση της, ε, του φίλου στον εμπορία ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Ε, εμπεριέχεται σε πολλές από τις συζητήσεις μας, σε διάφορες συγκυρίες, ε, και στο, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη για την καταπολέμηση της ε, άσκησης βίας κατά των γυναικών, των ε, νέων κτλ. Αυτή η ακρόαση έχει σαν στόχο να αναπτύξει και να προωθήσει και τις εργασίες για την εφαρμογή της οδηγίας του 2011-36 για την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων εδώ έχουμε δύο υπεύθυνου ε, εδώ στην ε, Επιτροπή. Έχουμε την εισηγήτρια την κυρία Βέρβερ και σαν ε, από πλευρά της Επιτροπής Γυναικών και ε, από την ε, Επιτροπή Ελευθεριών την κυρία Μπιόρκ. Είμαι σίγουρη ότι μαζί με τα άτομα τα οποία συμμετέχουν και στο πάνελ θα έχουμε μια αγώνιμη ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και όλα αυτά θα βελτιώσουν την γνώση μας και την συνειδητοποίηση των ε, γεγονότων. Η φιλετική βία και η σεματεμπορία των ανθρώπων είναι ένα, μια μάστιγα ε, και πιστεύω ότι χρειάζεται ε, μια εμπλοκή όλων των θεσμών και των κοινοτικών θεσμών ε, υπάρχουν διάφορες προοπτικές ε, και διαφορετικού, διαφορετικοί τομείς στους οποίους μπορούμε να εργαστούμε και ε, σε, αυτό το, σε αυτή την ακρόαση θα δούμε πολλές πτυχές του προβλήματος και θα το δούμε και από σφαιρική, θα διαμορφώσουμε μια σφαιρική άποψη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στους εισηγητές γιατί ε, θα ε, ε, ακούσουμε την κυρία Μπέρντερ και Μπιόρκ, που είναι οι συγγήτριες από τις επιτροπές μας, την Επιτροπή Γενικών και την Επιτροπή Ελευθεριών και ξεκινάμε με την κυρία Μπέρντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχουμε τους προσκεκλημένους ομιλητές να ακούσουμε. Είναι χαρά μου που είμαι η συγγήτρια όσον αφορά το την έκθεση εφαρμογής κατά του τράφικινγκ. Η ε, εμπορία των ανθρώπων είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει χρόνια και ε, ασχολούμαι με αυτό και στη χώρα μου και είναι μεγάλη ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να παρέμβει στην εργασία της Κομισιόν σε σχέση με το πρόγραμμα εφαρμογής, την έκθεση εφαρμογής. Λοιπόν, ο ορισμός ο οποίος χρησιμοποιεί στην οδηγία αντιτράφικινγκ είναι ε, ευρύς και προέρχεται και από προηγούμενες οδηγίες πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά για να απλουστεύσουμε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία βασικά θέματα. Ε, η εμπορία περιλαμβάνει την πράξη, τα μέσα και τον σκοπό τα μέσα είναι τα η αναγκαστική επιβολή αυτής της πράξης που αποδίδει κέρδος σε ένα άτομο το οποίο ελέγχει το θύμα. Τέλος, ο στόχος της ανθρώπινης εμπορίας είναι η εκμετάλλευση. Καμιά φορά αυτό μπορεί να εκλάβει πολλές ε, δραστηριότητες, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία κτλ. Και αν θέλετε αυτό υπάρχει, αυτός ο ορισμός συμβαδίζει με του ΟΗΕ. Αλλά υπάρχουν και διαφορετικοί ορισμοί στα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο σημαίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε πάντοτε να συνδυάσουμε τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι δεν περιλαμβάνουμε σε αυτή την έκθεση. Η εμπορία ανθρώπων, η σώματομπορία είναι ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο έχει σχέση και με την μεταναστευτική κρίση και την λαθρεμπορία ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν αυτούς που μεταφέρονται παράνομα, ε, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ΙΕ διαπιστώνει τρεις βασικές διαφορές. Ε, σεξουαλική εκμετάλλευση και ε, γενικά υπάρχει συνένεση σε αυτήν την παράνομη μεταφορά. Αρχική συνένεση η οποία βεβαίως έχει μετατραπεί σε αναγκαστική εκτέλεση. Το άρθρο 2, παράγραφος 4. Η συνένεση των θυμάτων στο τράφικινγκ δεν έχει καμία επιρροή ως προς τη διαπίστωση φτάνουν σε ένα προορισμό οι παράνομοι ε, λάθρομετανάστες ενώ ε, όταν έχουμε σώματεμπορία έχουμε συνεχή εκμετάλλευση. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν τράφικινγκ όταν μεταφέρεται το θύμα από ένα μέρος σε ένα άλλο, εσωτερικά σε ένα κράτος ή πέραν των συνόρων. Το τράφικινγκ, η εμπορία ανθρώπων, είναι κατάχρηση κατά του ανθρώπου. 69% όλων των εγγεγραμμένων θυμάτων του τράφικινγκ έχουν χρησιμοποιηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση. Από αυτό τον αριθμό το 95% είναι οι γυναίκες. Παρά την σπουδαιότητα της πορνείας μέσα στο πλαίσιο του τράφικινγκ πρέπει να διαχωρίσουμε ορισμένα πράγματα. Αυτή η έκθεση δεν δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε την προσέγγιση της πορνείας ειδικά έχουμε μεταφορά, ε, μάλλον εμπορία ανθρώπων, θύματα δηλαδή ανθρώπους που υφίστανται ένα έγκλημα και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι είναι που μας ενδιαφέρουν εδώ, δεν θέλουμε να ε, κρίνουμε τις συνθήκες της πορνείας γενικά. Δεν είναι αυτός ο στόχος δηλαδή. Η διάσταση του φίλου τώρα στην εμπορία ανθρώπων είναι σίγουρη. Έχουμε βέβαια εμπορία και αγοριών, αλλά η στατιστική δείχνει ότι τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και κορίτσια. Σύμφωνα με τη Eurostat, 80% των εγγεγραμμένων θυμάτων μεταξύ του 2010 και 2012 ήταν γυναίκες. Και αν και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Τα κράτη-μέλη τα οποία μπορέσαν να δώσουν περισσότερη ανάλυση των ηλικιών μας λένε ότι 70% ήταν μεταξύ 12 και 17 ετών και είχαμε και περιπτώσεις μεταξύ 2 και 11 ετών. μικρότερο ποσοστό βεβαίω. Οι στατιστικές δεν θα ανακλούν βέβαια την πραγματική κατάσταση και υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ καταχωρημένων περιπτώσεων και πραγματικότητας. Έχουμε το θέμα της ταυτοποίησης των ακτιμάτων του τράφικινγκ ανδρών και γυναικών. Αυτό έχει σχέση με τις διοκτικές αρχές και τις δικαστικές αρχές και τα θέματα της ταυτοποίησης. Αναφέρεται στην οδηγία ότι άνδρες και γυναίκες γίνεται εμπόριο ανδρών και γυναικών για διαφορετικούς λόγους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και υποστήριξη σε σχέση με το φύλλο. Εξειδικευμένα δηλαδή σε σχέση με το φύλλο. Πιστεύω ότι ορισμένα τμήματα της οδηγίας είναι πιο συγκεκριμένα από άλλα. Ε, στη γνωμοδίτηση της κυρίας Λό στην, ε, στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΑ θα ασχοληθούν με τα δικαστικά, τα νομικά εμείς θα ασχοληθούμε με τη νομική προστασία και την πρόληψη. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα και υπάρχουν διάφορα άρθρα τα οποία αναφέρονται στην προστασία των θυμάτων. Παρ' όλα αυτά τα θύματα της εμπορίας δεν έχουν καλή πρόσβαση προς τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα σαφές θέμα, με την ταυτοποίηση των θυμάτων, παρά την οδηγία ε, που ζητά μηχανισμούς για την πρόορη ταυτοποίηση και την υποστήριξη των θυμάτων. Οι υπηρεσίες για τα θύματα δεν χρηματοδοτούνται σωστά. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Και θα ήθελα να δω αν οι ομιλητέ μας έχουν κάτι να μας πούνε πώς μπορούμε να τα λύσουμε αυτά. Θα ήθελα ακόμη να ακούσω για τον επαναπατρισμό και την αποκατάσταση μακράς πνοής για τα θύματα. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές και ποιες είναι οι πολύ κακές πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά που θα μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπέρτερ. Κυρία Πιόρκο, εισηγήτρια, <coughs> συγγνώμη, ε, συντάκτρια γνωμοδότηση Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομη. Όπως είπε και η κυρία Μπέρντερ, η Επιτροπή μας ασχολείται με τα θέματα της επιβολής του νόμου, του ποινικού δικαίου. Θα έχουμε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Έχω ασχοληθεί με το θέμα της διακίνησης για πολλά χρόνια και πριν αναλάβω ως Ευρωβουλευτής. Το γυναικείο κίνημα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και το, να το γράψουμε στο θεματολογιό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που είναι αρμόδια καθήλυνη η Επιτροπή των Γυναικών γιατί μπορεί πιστεύω να προσφέρει τις πιο κατάλληλες λύσεις για την υλοποίηση και την εφαρμογή, την επιβολή του νόμου για την αντιμετώπιση διακίνησης εις βάρος των γυναικών. Προστασία όμως, δικαιώματα των γυναικών, των θυμάτων, πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε μεταξύ διαφορών μορφών ε, διακίνησης ή διακίνηση για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχει και πρέπει να έχει διαφορετική μεταχείριση είναι άλλο πράγμα από το γενικό όρο της διακίνησης ανθρώπων και άρα θα θέλαμε λύσεις τέτοιες από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Μπορεί κανείς να μην θέλει να υιοθετήσει διαφορετικές λύσεις προς την πολιτική τη σχετική με την πορνεία, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σχετική συζήτηση. Πρέπει να το παραδεχθούμε, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και πιστεύω ότι θα πρέπει ο στόχος μας να είναι όχι μόνο να προστατεύσουμε τα θύματα, αλλά και να αποτρέψουμε μελλοντικά την γένεση επιπλέον τέτοιων καταστάσεων και θυμάτων. Τι σημαίνει, τι είναι αυτός ο κλάδος, ποιες είναι οι συνθήκες εργασία, πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε οι συνθήκε διαβίωσης της εργασίας, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την, ε, την σώματεμπορία, ε, τι σημαίνει εκμετάλλευση για λόγους ε, σεξουαλικούς, για σεξουαλική εκμετάλλευση και τι σημαίνει και εκμετάλλευση για λόγους εργασιακούς. Αυτά νομίζω πρέπει να τα κοιτάξουμε μαζί. Περιμένω να ακούσω από τις και τον προσκεκλημένο μας ε, τις απόψεις του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπιόρκ. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας. Λοιπόν, για να οργανώσουμε το χρόνο να σας πω ότι θα σας δώσω 10 λεπτά στον καθένα. Θα πάρει πρώτα τον λόγο ο κύριος Γιώνα Χέντριξον, αστυνομικός επιθεωρητής από τη Στοκχόλμη. Ο κύριος Έριξον ασχολείται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορνεία και την εμπορία ανθρώπων από το 2008. Το 2013 μάλιστα απασχολείται πλήρως στη μονάδα για την πορνεία και είναι και μέλος ε, και της ε, ε, ειδικής ομάδας κατά της εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας. Πιστεύω ότι μπορεί να μας δώσει μια πολύτιμη συνεισφορά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χέντριξον που δεχθήκατε την πρόσκληση να συμμετάσχετε στην ακρόαση και σας δίνω αμέσως το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Και που με προσκαλέσατε. Και... Θα ήθελα να σημειώσω ξεκινώντας ότι η αστυνομική μου δουλειά έχει να κάνει με τόσο πολλές περιπτώσεις συλλήψεων για διακίνηση ανθρώπων. Έχω μόνο 10 λεπτά στη θέση μου. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω την κατάσταση και ελπίζω ότι μπορώ να δώσω και απαντήσεις ε, σε σχέση με κάποιες ε, τοποθετήσεις εσφαλμένες πιστεύω σε σχέση με την ε, Σουηδία. Έχουμε λοιπόν το θέμα της διακίνησης και της σωματεμπορίας. Σωματέμπορος είναι αυτός που κάνει να λειτουργεί το δίκτυο της διακίνησης. Έχουμε να κάνουμε με ε, αδικήματα που έχουν ε, σχέση με την ε, χρήση εκείνου δηλαδή που προσφέρει την υπηρεσία. Έχουμε να κάνουμε με αδικήματα που έχουν να κάνουν με εκμετάλλευση παιδιών, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Και την διακίνηση. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι της εργασίας μου. Όταν λοιπόν κάποιος προσπαθεί να κερδίσει χρήμα από την ε, σεξουαλική πράξη, πρόκειται για ένα πολύ ε, σοβαρό αδίκημα, διότι δεν είναι τόσο εύκολο να καταδικαστεί κανείς για τη διακίνηση, αλλά για την επικερδή προβολή, δηλαδή τη σωματεμπορία. Πολλέ είναι οι γυναίκες που έρχονται μέχρι τη χώρα μα ή που τις φέρνουν μέχρι τη χώρα μα οι διακινητές, αλλά μπορούμε να τους πιάσουμε κυρίως για την πώληση τη σεξουαλική ε, εξυπηρέτηση ως σωματέμποροι και ως αγοραστές βέβαια και ο αγοραστής σεξουαλικής υπηρεσίας γιατί ο παρέχον τη σεξουαλική υπηρεσία, η γυναίκα δηλαδή δεν ε, διώκεται. Ε, ο αγοραστής της σεξουαλικής πράξης, μπορεί να είναι και άντρας και γυναίκα βέβαια, γιατί ο νόμος μας είναι ουδέτερος, μπορεί να, δίνει, μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος πληρώνει όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε είδος, με αλκοόλ, με ναρκωτικά, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και βέβαια έχουμε ορίσει πρόστιμα. Το επιχείρημα μας είναι ότι με την νομοθεσία που έχουμε στο σουηδικό μοντέλο, το επιχειρήμα μάλλον που ακούγεται εις βάρος της νομοθεσίας μας είναι ότι με την νομοθεσία αυτή ε, σπρώχνεται προς την παρανομία όλο το ε, δίκτυο της ε, πώληση σεξουαλικών πράξεων. Βέβαια πολύ μεγάλη διάσταση παίρνει και το διαδίκτυο. Αυτό κοιτάμε και εμείς λοιπόν. Κοιτάμε για την ανείχνευση να ε, κάνουμε την αναζήτηση όπως τη κάνει και αυτός που αναζητεί να αγοράσει ε, σεξουαλικές υπηρεσίες και πάνω απ' όλα σε περίπτωση ανηλίκων. Βλέπετε εδώ στην οθόνη σας τις τιμές στο τιμολόγιο 150 ευρώ για 30 λεπτά με το κορίτσι αυτό. Να και το τηλέφωνο. Είναι απλά τα πράγματα. Παίρνει κανείς τηλέφωνο και απαντάει το κορίτσι αυτό το οποίο πωλείται σεξουαλικά και κλείνει κανείς ραντεβού. Αυτό έχω κάνει κι εγώ. Έχω πάρει τηλέφωνο, έχω κλείσει το ραντεβού, το κορίτσι μου στέλνει τη διεύθυνση και έτσι μπορώ να τη βρω. Και εκεί πάω βέβαια με την ομάδα μου, με τους συναδέλφους, στην διεύθυνση, χτυπάω το κουδίνο, λέω α εγώ είμαι έφτασα κτλ. Με καθοδηγεί στο ε, διαμέρισμα όπως έχει προβλεφθεί και βέβαια εγώ δεν μπορώ να πάω παραπέρα διότι είμαι αστυνομικό, αλλά ξέρω ποια είναι η ε, διεύθυνση που, πρέπει να, που εντοπίζεται έτσι και από αυτήν φτάνουμε στο υπόλοιπο δίκτυο. Εκεί λοιπόν, αφού δω το διαμέρισμα και τη διεύθυνση, βρίσκω μια δικαιολογία, έξαχασα το πορτοφόλι μου, δεν έχω λεφτά κτλ. και φεύγω. Και αρχίζει μετά η επιτήρηση του διαμερίσματος, η παρακολούθηση, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, γιατί ο καθένας μπαίνει ή βγαίνει είναι ύποπτος, ο σωματέμπορος και ξέρετε θα φτάσει κάποιος άντρας, πολλές φορές μάλιστα και περισσότεροι που κάνουν και ουρά και περιμένουμε να δούμε μπαίνουν στο διαμέρισμα που παρακολουθείτε. Μερικές φορές βάζουμε και κοριούς. Ακούμε τη διαπραγμάτευση για τις τιμές. Πολλές φορές παρακολουθούμε και τη σεξουαλική πράξη ακουστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να ε, ε, ξεκινήσουμε τη διαδικασία των διώξεων. Τους πιάνουμε την ώρα που βγαίνουν, τους κατάσχουμε το κοινικό τους, το, τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί θέλουμε τα στοιχεία, τα, την ηλεκτρονική αναζήτηση, τα SMS, τα mail που έχει στείλει, πώς έκρισε, δηλαδή ότι ακολούθησε την πορεία μιας διαφήμισης διαδικτυακής για να φτάσει στην αγορά της ε, υπηρεσίας της σεξουαλικής. Γίνεται βέβαια η ανάκριση αμέσως και οι περισσότεροι ομολόγουν ε, ευθέως ε, την πράξη τους γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν πολλές ψερότητες να αφωθούν αυτά φτάσουν στα δικαστήρια ομολογούν αμέσως πληρώνουν το πρόστιμο για να μην φτάσουν στα δικαστήρια μιλάμε με τα κορίτσια και η νομοθεσία που έχουμε δίνει άμεση πρόσβαση στις ε, κοπέλες αυτές οι οποίες είναι συχνά θύματα οργανωμένου εγκλήματος ε, σωματεμπόρων οι ίδιες ξέρουν ότι δεν έχουν διαπράξει έγκλημα και έτσι είναι ειλικρινείς μαζί μας, μας ε, μιλούν και έτσι μπορούμε και εμείς να τις πλησιάσουμε και να τις προσφέρουμε την βοήθεια που μπορεί να χρειάζονται, κοινωνική υποστήριξη. Κοινωνικός λειτουργός υπάρχει πάντα παρόν όταν συνομιλούμε μαζί τους και βέβαια προσπαθεί να τις ενθαρρύνει, να ξεφύγουν από την ε, πορνεία, να τους προσφέρει τα μέσα που θα χρειαστούν για να ξεφύγουν. Και πότε πότε βλέπουμε να πέφτει ο σπόρος και ένα-δύο χρόνια αργότερα που μπορεί να ξανασυναντήσουμε την ίδια κοπέλα, να τη δούμε σε καλύτερη κατάσταση, σε καλύτερες συνθήκες. Μιλάμε και με τους άντρες βέβαια για να τους εξηγήσουμε ότι βασικά χρηματοδοτούν το οργανωμένο έγκλημα και πολλοί δέχονται ή ζητούν ακόμη να ενταχθούν σε προγράμματα ε, ψυχοθεραπείας, σε ομάδες για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και να ξεφύγουν από αυτό το δίκτυο. Η νομοθεσία μας διευκολύνει λοιπόν πολύ. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη βία βάρος των γυναικών. 200 ανακρίσεις με γυναίκες ε, εκτεθειμένες στο δίκτυο της ε, πορνείας ή μάλλον ακροάσεις σχετικές με το δίκτυο της πορνείας ε, δείχνουν ότι δεν έχει επιδεινωθεί η κατάσταση για τις γυναίκες από την εισαγωγή αυτής της νομοθεσίας. Και μας λένε ότι είναι πολύ πιο ασφαλής, έχει περιοριστεί η βία εις βάρος τους ε, και πολλές φορές αποτρέπεται και ο υποψήφιος πελάτης γιατί ξέρουν ότι μπορεί να διωχθεί ως αγοραστής της σεξουαλικής υπηρεσίας εμεί μπορούμε να παρακολουθούμε και να έχουμε επικοινωνία με τι γυναίκε να ξέρουμε τι διευθύνσεις του να, να συνομιλούμε μαζί του και να του προσφέρουμε βοήθεια. Επίσης, ε, άρα λοιπόν ε, καταραίει το επιχείρημα ότι με την νομοθεσία αυτή έχει αυξηθεί η βία εις βάρος των γυναικών. Το ίδιο και με το ότι υποτίθεται πως είναι παράνομες οι παρακολουθήσεις, η κορία κτλ. Όχι, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τους υπόπτους και να έχουμε αποτελεσματική δράση. Ε, βλέπουμε ότι η νομοθεσία αυτή δηλαδή έχει αλλάξει και τις νοοτροπίες στην ε, Σουηδία. Πια δεν θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή η χρήση της υπηρεσίας της ε, πορνείας. Είναι καταδικαστέα περισσότερο κοινωνικά και αντίστροφα οι γυναίκες μας μιλάνε πολύ πιο άνετα, πολύ πιο ελεύθερα. Έχουμε καταφέρει δηλαδή ένα σοβαρό πλήγμα στην αγορά την ίδια. Έχουμε αντιστρέψει την εικόνα της αγοράς ε, των σεξουαλικών υπηρεσιών, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τις γυναίκες. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι και άλλες χώρες θα δουν θετικές εξελίξεις αν υιοθετήσουν το μοντέλο, το μοντέλο μας. Και οι τιμές ακόμα έχουν ε, αλλάξει, έχουν <coughs> αυξηθεί, γιατί φοβούνται οι πελάτες την ε, καταγγελία και άρα πληρώνουν την, την τιμή που ε, ζητείτε και ναι, δεν θα πούμε ότι πρόκειται για γυναίκες ευτυχισμένες ε, εργάτριες ε, της γενετήσιας ε, συνέβρεσης οι οποίες χαίρονται να πάνε να προσφέρουν το κορμί τους. Όχι, πολλές φορές είναι κοπέλες φτωχές σε δύσκολες συνθήκες που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. Και άρα θέλουμε να τις βοηθήσουμε γι' αυτό και σημειώνω τα κλειδιά της επιτυχίας μας ότι ποινικοποιείται η αγορά της σεξουαλικής υπηρεσίας. Έχουμε σοβαρές ε, κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Έχουμε καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και βέβαια διατίθεται και σοβαρή ε, αστυνομική ε, δύναμη διαθέσιμη για να καταπολεμηθεί το σωματεμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, señor ευχαριστώ πολύ, κύριε επιβεβαίωσα ότι αυτό που είπα στην αρχή ήταν πολύτιμη συνεισφορά σας εφόσον εργάζεστε επί τόπου και βλέπετε καθημερινά ε, αυτά τα ζητήματα. Είδαμε και εμείς λοιπόν, ε, πήραμε μια γεύση της δουλειάς που γίνεται επί τόπου καθημερινά και είναι πολύ θετικό αυτό γιατί έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε πολλές γυναίκες ε, να βγουν από επονίδιστες καταστάσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρέιτσελ Μοράν συγγραφέα και μέλος της οργάνωσης Space International. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο που μιλά ακριβώς για αυτό το θέμα της ε, πορνείας. Η οργάνωση Space International, στην οποία ε, ανήκει, δίνει φωνή στις γυναίκες οι οποίες έχουν βιώσει κακοποίηση, είναι θύματα ή μάλλον εργάζονται ε, ως ιερόβλης και τα λοιπά. Ε, θα μας δώσει λοιπόν και η κυρία Μωράν την άποψή της. Ε, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και σας δίνω μέσα στο λόγο. Ναι, ναι. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να διορθώσω ε, την παρανόηση στη μετάφραση στον υπότιτλο του βιβλίου μου. Πρόκειται για το, τη διαδρομή μου μέσω της πορνείας. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει εδώ και καιρό είναι ότι η πορνεία ε, δεν είναι μία εργασία, είναι μία κατάχρηση. Και μπορώ να σας, πω, να σας το πω αυτό ε, περνώντα 7 χρόνια μέσα στο πλαίσιο, ε, πολλά χρόνια γράφοντας, πολλά χρόνια επεξεργαζόμενοι τις απόψεις μου και τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζομαι με γυναίκες εντός και εκτός του πλαισίου του Space International. Η πορνεία λοιπόν υπήρξε κομμάτι της ζωής μου για 25 χρόνια με τον ένα τρόπο και τον άλλο. Συνεπώς μπορώ να πω ότι έχω καθήκον και υποχρέωση να πω ότι ποτέ εδώ ή αλλού δεν θα ισχυρίσω, δεν θα ισχυριστώ ότι η εμπορία, η σωματεμπορία είναι διαφορετική από την πορνεία. Διότι η σώματα το trafficking, είναι ένας τρόπος μετακίνησης είτε στο εσωτερικό χωρών, είτε διεθνώς, είτε σε όλη Η πορνεία είναι η κατάληξη της εμπορίας για σεξ. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν δεν υπήρχε πορνεία, δεν θα υπήρχε και η εμπορία ανθρώπων για το σεξ. Έχω συναντήσει γυναίκες που υπήρξαν ε, θύματα σωματεμπόρων με την νομική έννοια. Και συγκεκριμένα έχω μια γυναίκα που συνάντησα από τη, στη χώρα μου και είναι κλασική περίπτωση όσον αφορά την εμπορία για το σεξ. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και διαφορετικοί τύποι καταναγκασμού η γυναίκα αυτή κυριολεκτικά τη σύρανε από τα μαλλιά και τη βάλανε σε ένα φορτηγό στο Λονδίνο και την πήγαν στο αεροδρόμιο αφού ε, πήραν το, ε, το διαβατήριό της και πέρασε τα χρόνια της σε οίκους ανοχής της Ιρλανδίας για πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτό έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για trafficking, για σεξ. Λοιπόν, από την εμπειρία που είχα και από όσα είδα στις ζωές πολλών γυναικών στα 7 χρόνια στα οποία ενεπλάκην εγώ η ίδια, μπορώ να σας πω ότι ο καταναγκασμός είναι μέσα στο πλαίσιο εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει πράγμα σαν αυτό που λέμε ε, μια ευτυχής γυναίκα η οποία ελεύθερα συμμετέχει στην πορνεία αποκλειστικά ε, χωρίς κανέναν καταναγκασμό. Δεν υπάρχει τέτοια γυναίκα. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε εδώ είναι ότι σε αυτή τη ε, γη αν τη θεωρήσουμε σαν μια σφαίρα αντί να κοιτάμε τους εαυτούς μας και είναι το πιο φυσικό που κάνουμε να κοιτάμε τον εαυτό μας. Θα βλέπαμε αν κοιτούσαμε τη σφαίρα ότι υπερέχει σαφέστατα ε, υπερέχουν ε, σαφέστατα οι γυναίκες που είναι από φτωχό περιβάλλον, έγχρωμες και στην Ιρλανδία όπου μεγάλωσα μπορώ να σας πω ότι οι γυναίκες που μπήκαν στην πορνεία ουσιαστικά μπήκαν σε αυτήν όταν ήταν πολύ νέες κορίτσια, εγώ μπήκα στα 15 και 15, 16, 17 είναι οι ηλικίες εισόδου. Έχουμε λοιπόν το κοινωνικό σύστημα φροντίδας, ε, το οποίο όμως δεν είναι αποτελεσματικό και δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι το τράφικινγκ για το σεξ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ε, σε ταινίε και σε κάπου 10-15% του συνολικού εμπορίου του σεξ και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι ε, ευτυχισμένες γυναίκες οι οποίες ελεύθερα έχουν επιλέξει την πορνεία. Λοιπόν, Έχω δει πάρα πολλά πράγματα στην πορνεία και ε, ε, πραγματικά ελεύθερη επιλογή δεν υπάρχει. Ελεύθερη επιλογή είναι κάτι το οποίο μπορείς να μετρήσεις σε σχέση με κάτι βιώσιμο. Και μπορώ να σας πω ότι με έχει κουράσει το να πηγαίνω σε διάφορα μέρη και να μου λένε ότι η εμπορία για το σεξ και η πορνεία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς και αληθινοί αν πρόκειται να μιλήσουμε για την πορνεία. Η πορνεία είναι η χρήση του σώματος ενός κοριτσιού ή μιας γυναίκας από έναν άντρα συνήθως και όταν μιλάμε για τη διάσταση του φίλου για την εμπορία θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Χαίρομαι ακόμη που βρίσκομαι εδώ με τον αξιωματικό Χέντριξον, διότι η σουηδική αστυνομία τα καταφέρνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη αστυνομία έχω συναντήσει στον κόσμο και χρειάζεται να εμπνευστούμε από όσα γίνονται στη Σουηδία. Τώρα, δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θέλω να καλύψω τον χρόνο άλλων ομιλητών. Θα σας πω μερικές σκέψεις σύντομα σε σχέση με τις ενδεχόμενες λύσεις στους πολιτικούς κύκλους όπως συζητούνται. Η πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Ζηλανδία από ποινικοποίηση. Αυτό είναι το μοντέλο της. Θα ήταν σχεδόν διασκεδαστικό για μένα, πρέπει να σας πω. Είναι στρεβλό, δηλαδή είναι κάπως διαφορετικό από τα πρότυπα νομιμοποίησης της Γερμανίας, της, Αυστραλίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας κτλ. Διότι οι νέες γυναίκες ε, στη Νέα Ζηλανδία μου λένε ότι πρόκειται για ακριβώς παρόμοιο πράγμα με αυτό που συμβαίνει στις χώρες που μόλις ανέφερα. Και θα ήθελα να, να μου πείτε ε, σε ποιο πλανέτη ότι πλανήτη ζούμε θεωρώντας ότι η νομιμοποίηση ή η αποποινικοποίηση καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Προημερών συνάντησα μια άλλη κοπέλα από τη Νέα Ζηλανδία. Αυτή η συγκεκριμένη βγήκε από την πορνεία, δεν έχει πολύ χρόνο και αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο στις συζητήσεις με τις Νέο Ζηλανδές εντυπωσιάζομαι από το εξή γεγονός. Όταν εξηγώ ότι στη ΣΥΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη ε, εκείνοι που είναι πολιτικοί αντίπαλοι ε, δίδουν παραδείγματα σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση νομοθετικά, εντυπωσιάζουν όταν τους μιλάω γι' αυτό τι οι Νέο Ζηλανδές. Θα σας πω πώς λειτουργεί το σύστημα στην πραγματικότητα. Αποποινικοποίηση ή νομιμοποίηση. Αν αποποινικοποιήσετε τους προαγωγούς, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, διότι καλά περνάνε εν πάση περιπτώσει. Έχω ένα παράδειγμα να σας δώσω. Νόμιζα ότι τα ξέρα όλα, αλλά συνεχώς υπάρχει και κάτι καινούριο που εμφανίζεται δεν υπάρχει τέλος στην ασθένεια του διεθνούς εμπορίου σεξ. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάθε τόσο κάτι καινούριο που λες Θεέ μου. Αυτή λοιπόν η νέα κοπέλα μου εξήγησε ότι σε ένα από τα πορνεία στα οποία δούλεψε, μιλούσε πολύ γρήγορα και σχεδόν δεν το κατάλαβα την πρώτη φορά, μου είπε «Θεέ μου, δεν έχουν καν σεντόνια εκεί» και είπα τι εννοεί. και μου λέει είναι ένα πορνείο που λειτουργεί 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, άνδρες και γυναίκες και δεν μπορείτε να έχετε ε, σε δόντια, θα έπρεπε να αλλάζουν συνέχεια. Οπότε έχουν ειδικά στρώματα ε, πλαστικοποιημένα και με ένα σπρέι τα καθαρίζεται αυτά, τα απολυμένεται. Λοιπόν, οι άνθρωποι αν δεν καταλαβαίνουν τη φρίκη της πορνείας, ίσως δεν καταλαβαίνουν και αυτό το οποίο με ενοχλεί προσωπικά τόσο πολύ. Αυτή η γυναίκα λοιπόν μιλάει απλά για το ότι δεν υπάρχουν σεντόνια και, και θα αναρωτιόσαστε γιατί με απασχολεί αυτό. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η πορνεία όταν αποποινικοποιείται, οι εκμεταλλευτές δηλαδή και οι πράξεις τους αποποινικοποιούνται ε, δημιουργεί πρόβλημα στις γυναίκες. Τι έχει συμβεί. Έχουν γίνει απάνθρωπες οι συνθήκες. Θα μπορούσαν ε, να έχουμε τις γυναίκες να παρουσιάζονται σε ένα κινούμενο ημάντα. Αυτό συμβαίνει στη Νέα Ζηλανδία και σε άλλες χώρες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται. Μας λένε ότι αυτό είναι το τέλειο μοντέλο. Λοιπόν, εγώ έχω πολλά να πω γι' αυτό, προτού σιωπήσω και το αφήσω να προχωρήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κανείς είναι μέλος της Άμνεστη. Λοιπόν, αν ήσασταν θα σας ρωτούσα γιατί ο Ντόγκλος Φόξ, Βρετανός προαγωγός ε, προχώρησε σε αυτή την πρόταση. Πρώτη σημαντική ερώτηση. Η Άμνηστη ε, έθεσε αυτό το θέμα στη Βόρεια Ιρλανδία το 2014. Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί το παγκόσμιο δίκτυο προσφέρει απόψεις στο δίκτυο όταν ο Αλεξάνδρ Γκίλ και η μια κυρία ήταν υπεύθυνε για το εμπόριο στο Μεξικό. Λοιπόν, μιλάμε εδώ για την διάσταση του φύλου του εμπορίου χωρίς να μιλήσουμε για τη συμβολή των προμηθευτών. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Muchísimas eh, eh, ευχαριστώ πολύ, κυρία Μωράν, που μα μεταφέρατε με τα λόγια σα. Ε, Εικόνε και ζητήματα που πολλέ φορέ μα απασχολούν στην Επιτροπή μα αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη. Όχι τόσο ίσω ω πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών αλλά εκ του προσωπικού μιλώντα πραγματικά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να γίνεται ε, διάκριση μεταξύ εμπορίας ανθρώπων και πορνείας, ε, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για να είναι πιο διαδραστικό και συμμετοχικό τώρα το πλαίσιο, θα δώσω το λόγο στις κοιότητες εισηγητρίες για τις δύο εκθέσεις των δύο ομάδων. Η κυρία Κοράτσα, καταρχάς από το ΕΛΚ, έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Η ομιλήτρια δεν ακούγεται, είναι χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται ακόμη, το μικρόφωνο δεν έχει ανάψει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω πως ε, με συγκίνησαν πολύ οι περιγραφές ε, των φρικαλαιότητων στις οποίες εκτιθέτει οι γυναίκες, ε, θύματα της εκμετάλλευσης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης που μας δώσατε και χαίρομαι που είπατε πολύ συγκεκριμένο ότι πρόκειται για παιδιά συχνά, κορίτσια μικρά, που είναι, πέφτουν θύματα αυτών των κυκλωμάτων, όλο και περισσότερα. Και βέβαια είναι τα πιο ευάλωτα. Όλο και περισσότερα και κάθε ιστορία είναι μια τραγωδία. Πολλές φορές είπατε και εσείς ότι δεν υπάρχουν επιλογές και τα οδηγεί η φτώχεια σε αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι που δίνει κάποιες λύσεις, έστω κάποιες λύσεις, η Σουηδική νομοθεσία και είναι αποτελεσματική. Βεβαίως θα ήθελα να αναφερθώ και στον προφανή σύνδεσμο μεταξύ ε, σωματεμπορίας ε, και μετανάστευσης. Έχω επισκεφθεί την Λαμπεντούσα, την νότια οχθή της ε, Μεσογείου, στο Μποντρούμ, την άλλη καρνισό της Τουρκίας, ε, έχω συνομιλήσει με ομάδα γυναικών που προσπαθούν κάθε βράδυ ε, γυρνώντας ε, στους δρόμους να εντοπίσουν γυναίκες που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Έχω, έχω συνομιλήσει με την οργάνωση της Λαμπετούζα που αντίστοιχα προσπαθεί να εντοπίσει τα δίκτυα διακίνησης γυναικών Φερρυπίν από την Ιγυρία, γνωστό δίκτυο και επίσης ένα πολύ καλό ε, σεμινάριο που διοργανώθηκε από την συντονίστρια για την καταπολέμηση της ε, ε, λαφροδιακίνησης ανθρώπων σωματεμπορίας και όλοι μας λένε το ίδιο πράγμα, ότι τα δίκτυα είναι γνωστά. Οι διακινητές είναι γνωστοί, ξέρουν τα ονόματά τους ακόμη. Και όταν φτάνει η ώρα να παραμεθούν στη δικαιοσύνη, στη Σικελία δεν υπάρχουν αρκετά αποδει αποδεικτικά στοιχεία, γιατί οι φωτογραφίες τους δεν αρκούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον των δικαστηρίων. Και έχουν ε, τεράστιο αίσθημα απογοήτευσης και ματέωσης, διότι με όλες τις προσπαθίες τους, ακόμα και με μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δουλεύουν, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν καταδίκες από τα δικαστήρια αφού τα αποδεικτικά του στοιχεία δεν αρκούν. Αυτό λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση των πόρων, των, των ανακριτικών εξουσιών για τη Eurojust, για τη Europol και εσάς ιδιαίτερα ως ε, αστυνομικό επιθεωρητή. Θέλω να σας ρωτήσω, η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τρίτες χώρες, με χώρες ε, ε, διακίνησης η διέλευση καλύτερα, όπου πάντα δεν είναι εύκολη η επικοινωνία και η τελική δεδομένων. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς είμαι και σκιώδης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πώς μπορούμε εμείς να παροτρύνουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη βελτίωση αυτών των συνοδικών με τις οποίες εργάζεστε και πώς επίσης μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με το δικαστικό, με το σύστημα της απονομής της δικαιοσύνης, οι ε, επιτυχίες της καταδίκες. Και βεβαίως η χρηματοδότηση αυτής της διακίνησης είναι τεράστια τα κέρδη που αποφέρει για το οργανωμένο έγκλημα, δισεκατομμύρια ευρώ σε κέρδη, πώς μπορούμε να ανοιχνεύσουμε, να παρακολουθήσουμε και να δώσουμε και τα κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ε, παταχθεί ατιμορρησία και να διαλυθούν αυτά τα δίκτυα. Ευχαριστώ πολύ, Κοράτσα. Κύριε Χάνιμπολ, εκ μέρου των Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τι ομιλητρίε και του ομιλητέ. Είναι πολύ καλό που συζητούμε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί κανείς να εξαντλήσει αυτό το θέμα, τουλάχιστον αυτή την η προσωπική μου άποψη και χαίρομαι που μας δίνετε μια ακόμη ευκαιρία να το κάνουμε και για τις γυναίκες ε, πραγματικά είναι ζήτημα που αφορά τις γυναίκες κυρίως, είναι ε, και θέμα φίλου. Ε, ξέρω πώς το συζητάμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον έξω από εδώ αντιλαμβάνεται κανείς ακριβώς τη διάσταση του προβλήματος. Ίσως όχι στη Σουηδή γιατί αλλάζουν οι στάσεις και οι συμπεριφορές, αλλά σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες η πορνή δεν θεωρείται κάτι απλά που πάντοτε υπήρχε ε, μαζί μας, αλλά σαν να υπάρχει αυτοδικαίως κατά κάποιο τρόπο. Ε, και πολλές φορές ε, είναι φρικτό αυτό, αλλά συζητείται και αστεί, και αστεία πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς κάπως τα πράγματα, αρχίζοντας ίσως να συζητούμε ως γυναίκες το ζήτημα αυτό με σοβαρότητα και σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτή η διασύνδεση των δύο φαινομένων να βρει κοινή γνώμη, δηλαδή ε, πορνείας και σωματεμπορίας. Ε, Προσωπό το Λονδίνο, που γνωρίζετε, είναι προορισμός και είναι πολύ σημαντικό όπου και από όπου και αν προερχόμαστε βέβαια, αλλά αν προερχόμαστε από μέρη όπου υπάρχει ζήτημα με την εμπορία ανθρώπων, να συνεχίσουμε να ε, κάνουμε εκστρατεία πληροφόρησης. Ε, και να συνδέουμε την πονία, τη διακίνηση ανθρώπων και ε, όλο το ζήτημα αυτό, αυτό του φίλου και πρέπει να σπάσουμε όλους τους μύθους που υπάρχουν. Άκουσα και κάποια που επιβεβαιώνουν ε, κάποιες υποψίες που είχα. Η οργάνωση είναι πολύ σημαντική, τη σέβονται πολύ και το ψήφισμα ξέρω επίση ότι δημιούργησε κάποια προβλήματα. Εμείς πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθούμε όσο μπορούμε περισσότερο το σουηδικό μοντέλο, που βέβαια ε, και με ψήφισμα στο Κοινοβούλιο ε, προωθούμε και εγώ προσωπικά είμαι προσλημμένη σε αυτή την πολιτική. Επαναλαμβάνω, όσοι και όσε ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία πληροφόρηση και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα πιο πέρα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πού μπορεί ε, να βοηθήσει για να υλοποιηθούν κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα μπορούμε να το προωθήσουμε ακόμη περισσότερο. Και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας πάνω στο θέμα της εμπόριας ανθρώπου. Και ο, η μείωση της ζήτησης είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Είναι σημείο κλειδί. Και δεν υπήρξε μέχρι στιγμής άλλο νομοθέτημα που μειώνει την ε, ε, ζήτηση, αλλά παρά το σφιδικό αυτό μοντέλο και ελπίζω να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να πετύχουμε περισσότερα και ως κοινοβούλιο. Γιατί το κοινοβούλιο έχει ε, αποφασιστικές πολιτικές για αυτά τα θέματα. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη μετανάστευση και να τα συσχετίσουμε αυτά τα ζητήματα. Μάλλον θα αναλάβω τη σύνταξη έκθεση πρωτοβουλίας επιτροπής μας για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι και αυτή η πτυχή είναι μια ακόμη διάσταση του όλου προβλήματος. Όταν έχουμε μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων, πάντα ε, τα φαινόμενα εκμετάλλευσης και κακοποίησης ε, αυξάνονται και πρέπει να το δούμε και αυτό πιστεύω. Ίσως έτσι έχουμε ένα πιο γενικό πλαίσιο για να θέσουμε και τα άλλα ζητήματα που είναι και ίσως πιο μακροπρόθεσμα και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις εθνικές νοοτροπίες, τάσεις και συμπεριφορές. Πολλά έχουμε να κάνουμε πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές του πάνελ και ελπίζω μετά από αυτήν την ε, ακρόαση Σίγουρα δεν έχουμε παραιτηθεί ποτέ στην Επιτροπή των Γυναικών, αλλά ελπίζω η σημερινή μέρα να μας δώσει ακόμη περισσότερα εφόδια και πυρομαχικά για να κάνουμε πιο πολλές προτάσεις και να πάρουμε πιο πολλές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ο κύριος ε, Έριξον ή η κυρία Μωράν θα θέλαν να κάνουν ε, κάποιες ε, παρατηρήσεις, αν έχουν εκφράσουν κάποιες σκέψεις τους μετά από όσα άκουσαν. Α, όχι, πριν από αυτό όμως η κυρία Μπέρντερ θέλει να κανουν καποιες παρατηρησεις αν εχουν εκφρασουν καποιες σκεψεις τους μετα απο οσα ακουσαν α πριν απο αυτο ομως η κυρια μπερντερ θελει να παρει το λόγο. Πριν... Ναι, πριν πάμε στις απαντήσεις. Έχω μια δύο ερωτήσεις ακόμα. Ο σύνδεσμος μεταξύ πορνείας και δεν το αρνούμε όταν μιλούμε για την ε, σωματεμπορία. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή η πορνεία δεν θα υπήρχε η σωματεμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση. Αλλά νομίζω ότι η λαθροδιακίνηση ανθρώπων ξεπερνάει την πορνεία. Και όπως είπα στην αρχή δεν θέλω να εκφέρω ε, ηθικές αξιολογήσεις για την πορνεία. Και όλο αυτό το ζήτημα της, ε, του εξαναγκασμού, και της πορνείας. Με ενδιαφέρει, έχω δει και ένα σεμινάριο στο Λονδίνο με εκπροσώπους οργανώσεων ιερόδουλων που μας έλεγαν ότι όλα είναι πολύ ωραία σε αυτόν τον κόσμο και ότι ξυπνάει κανείς, ε, είναι 15 ετών και αποφασίζει να πάει να ε, πουλήσει έρωτα. Ε, σαν να ήταν μια επιλογή σταδιοδρομίας για τα νεαρά κορίτσια. Επιπλέον όμως αυτό να υπάρχει και η σωματεμπορία δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Για μια διευκρίνηση όμως σε σχέση με τη Σουηδία. Ε, έχει αλλάξει όπως είπατε και η νοοτροπία σε όλη την κοινωνία στη Σουηδία για το τι συμβαίνει μεταξύ ανδρών και γυναικών και τι σημαίνει το να αγοράζει κανείς την πρόσβαση στο κορμί κάποιου άλλου. Αλλά τι κάνουν Εκείνοι που είναι στην πρώτη γραμμή, οι αξιωματούχοι που εργάζονται, τι κάνουν τα δικαστήρια, αφού έγινε λόγος για την ατιμορρησία. Όταν ε, συνομιλείτε με τι ε, κοπέλε μπορούν να σα δώσουν στοιχεία και να αποκαλύψουν ότι είναι θύματα λαθρεμπορίου, σωματεμπορίας. Μπορούν να δώσουν τα στοιχεία αυτά και μπορούν από εκεί να ξεκινήσουν την ε, δράση του οι αρχέ χωρί να κινδυνεύουν οι κοπέλε, να βρεθούν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση μόλι γυρίσετε την πλάτη σα και νομίζετε ότι πράγματι έχει περιοριστεί η λαθροδιακίνηση στην Σουηδία ή απλώς την έχετε σπρώξει σε κάποια άλλη χώρα. Και ναι, ευχαριστώ για όσα ακούστηκαν. Όντω είναι πολύ δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ της διακίνησης και του εισπορνίας. Αλλά η χρήση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράνομο να ε, χρησιμοποιήσει κανείς τις υπηρεσίες κάποιου για τον οποίο γνωρίζει ότι έχει πέσει θέμα, θέμα διακίνησης. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν μια κοπέλα να λέει, λέει να ενημερώνει τον πελάτη ότι χρειάζεται βοήθεια γιατί είναι θέμα διακίνησης κάποιου δικτύου σωματεμπορίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Η Μέρη αναφέρθηκε στο Λονδίνο. Εμείς είχαμε στην Οξφόρδη μια ε, ένα μεγάλο σκάνδαλο ε, που αφορούσε πολλά κορίτσια που όταν πια δεν προστάτευαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτου έπεσαν στην πορνεία και στην εκμετάλλευση σεξουαλική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε ότι αν δεν υπήρχε η πορνεία δεν θα υπήρχε εμπόριο σεξουαλικών υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη και νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση. Βλέπω, καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι υπάρχει μεγάλο κομμάτι εξαναγκασμού σε στην υπόθεση τη πορνεία. Αλλά πώ από τα κορίτσια αυτά είναι θύματα δια, λάθρο διακίνηση ή σωματεμπορία, το έχετε βρει αυτό. πώ είναι αυτά δηλαδή, τα οποία διακίνησαν κάποια δίκτυα και δεν είναι απλώ ένα κορίτσι τη γειτονιά που δεν είχε λεφτά και αναγκάστηκε. Άλλες δύο συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στο πάνελ. κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία σύντομη ερώτηση. Να ευχαριστήσω και τους δυο σας ε, για, ε, ε, για την εξαιρετική συνεισφορά σας. Μας δώσετε να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Απλώς θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χένριξον πώς Είπατε μάλλον ότι είναι χρήσιμο να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκριμα και τη σωματεμπορία και η σουδική νομοθεσία προβλέπει ε, κάτι τέτοιο. Πώς το κάνετε όμως, τι σημαίνει συγκεκριμένα δηλαδή αυτό. σε σχέση και σε σύγκριση με τις δράσεις της αστυνομία σε άλλες χώρες που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Επίσης, για αυτούς που θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω, όπως εγώ παραδείγματος χάρη, οργανώνουμε ένα εργαστήρι στις μία η ώρα, επαναλαμβάνω, όπου ε, θα ενημερωθούμε για το τι γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες. Θα ενημερωθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Η κυρία Γουίντσμπερκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο, ευχαριστώ και για τις παρεμβάσεις που ακούσαμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Χαίρομαι που ακούμε για αυτό το σουηδικό μοντέλο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Γιώνας. Για τους πόρους, έχετε επαρκείς πόρους, ε, αυτούς που χρειάζεστε τουλάχιστον γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κύμα, μια ροή, μεγάλη ροή ανθρώπων που φτάνουν στη Σουηδία και αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα ε, είναι μεγαλύτερο τώρα. Ε, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ μας είπε ότι ξέρουμε και τα ονόματα των σωματεμπόρων και των διακινητών ε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι διότι αυξηθεί και ο αριθμός των ανθρώπων που θα έρθουν στην, στη Σουηδία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Έχω την αίσθηση ότι η αστυνομία χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Αυτό ισχύει στη Σουηδία νομίζω. Επίσης είπατε ότι θέλετε να κάνουμε την αγορά λιγότερο ελκυστική. Αλήθεια είναι αυτό, διότι ε, θα στραφείτε και εναντίον των αγοραστών. Όντως κάνετε την αγορά λιγότερο ελκυστική. Αλλά εγώ σκέφτομαι και τις γυναίκες Μήπως θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες περισσότερο με τη δημιουργία καταφυγίων, ε, ε, κέντρων υποδοχής. Ε, θεωρείτε ότι βοηθάμε αρκετά τις γυναίκες ώστε να μην επιστρέψουν στην ίδια κατάσταση μετά. Ακούσαμε ότι ας πούμε πολλές φορές οι γυναίκες μετά από μερικά χρόνια ξαεπιστρέφουν. Κυρία Κοράτσα Μπίλντερ. Ήθελα να κάνω, να, θέλω να καταστήσω σαφέ, συγγνώμη, ότι μιλάμε για καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων, των εγκληματιών, που, ε, που εκμεταλλεύονται τους ε, μετανάστες. Δεν ε, καταπολεμούμε την μετανάστευση. Εμείς συζητήσαμε συμπληρωματικούς πόρους, συμπληρωματικές ενισχύσεις, αν θέλετε, της Frontex και των άλλων υπηρεσιών που δρούν στην Μεσόγειο, την, αυτούς που ελέγχουν τα σύνορα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους μετανάστες και κυρίως τα παιδιά των μεταναστών. Δεν λέμε να κρατήσουμε τους μετανάστες έξω από την Ευρώπη, αλλά όταν μπουν στην Ευρώπη να μην πέσουν στα δίκτυα των διακινητών. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος, ε, ε, η κυρία Μωράνη, ο κύριος Χέντριξον να θέλουν να πάρουν το λόγο. Α, είναι λίγο καινούργια αυτή η διαδικασία. Για μένα έχω πάρει σημειώσει, θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Σε ό,τι αφορά όσα είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτα, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, πάντοτε θέλουμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα και φυσικά χρειαζόμαστε πάντοτε περισσότερα μέσα και πόρου. Είναι προφανέ αυτό. Αυτό που θα ήθελα εγώ προσωπικά θα ήταν ε, σε επίπεδο κεντρική οργάνωση να έχουμε κάποιε απαιτήσει για το πώ πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Αλλιώ ε, η ε, ε, αστυνομία θα λέει ότι δεν έχουμε πόρου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε όλα αυτά και τα βάζουμε κατά το χαλί τελικά τα προβλήματα. Αλλά έτσι θα έχουμε 200 λιγότερες συλλήψεις τη με άνδρες που αγοράζουν σεξ. Και βέβαια τα προβλήματα δεν είναι μόνο στο χαρτί, είναι πιο σοβαρά. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσει στις άλλε χώρε ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση ω προ αυτό το φαινόμενο. Γιατί πιστεύω ότι περισσότερες περισσότερε από τι γυναίκε που είναι αντικείμενο εκμετάλλευση είναι αντικείμενο εκμετάλλευση γιατί όπως είπε η Ρέιτσελ δεν έχουν άλλη επιλογή. Οι δε εκμεταλλευτές είναι οργανωμένοι από δική τους πλευρά εργάζονται ε, κεντρικά, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και έχουν και πάρα πολύ ε, χρήμα στη διάθεσή τους. Πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι βλέπετε, παραδείγματο χάρη, ε, στην περίπτωση όπλων και μπορούν να καλύπτουν ε, και τα κενά και τα παραθυράκια που έχουμε στο σύστημα πρόληψης. Εμείς στην Σουηδία, στη το έχουμε αυτό το σύστημα ε, ανείχνευση εντοπισμού, αλλά δεν υπάρχει παντού αυτό. Πρέπει λοιπόν να, να δούμε τι γίνεται αλλού και να φροντίσουμε να κόψουμε ε, να, αυτά τα φαινόμενα από τη ρίζα και σε άλλες ε, χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, πού είναι το χρήμα και πολλές επιχειρήσεις, ξέρετε, στα Σουηδία σταματάνε στα σύνορα. Ε, στη Ρουμανία, για παράδειγμα, πηγαίνουν κάποια κονδύλια, κάποια χρήματα και μένουν εκεί. Ε, εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε πέρα από τα σχετικά σύνορα. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της αστυνομίας έχουμε ένα γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχουμε και μακρά κληρονομιά και παράδοση στη Σουηδία σε ό,τι αφορά τις ίσες ευκαιρίες, σε ό,τι αφορά διάφορους τομείς ε, τεχνογνωσίας, ε, εμπειρογνωσίνη. Και φυσικά αν κάποιος προσληφθεί για να εργαστεί σε αυτό το τομέα θα προσληφθεί με βάση την εμπειρία του ή της. Βέβαια πάντοτε επενδύουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία του προσωπικού μας, ε, την εκπαίδευσή του. Μέχρι στιγμής πάντως καλά είναι τα αποτελέσματα. Τώρα, ε, ό,τι αφορά το κατά πόσο τα κορίτσια ε, γυναίκες ε, νιώθουν ελεύθερες να μας μιλήσουν. Μας μιλούν. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν και το αντιλαμβάνονται εκ των μυστέρων. Δηλαδή, μας λένε πολλές φορές δεν μπορούσα να σας το πω δύο χρόνια πριν, αλλά αποβίωσε ο πατέρας μου πριν δύο χρόνια στη Γερμανία και τώρα μπορώ να σας μιλήσω για το παρελθόν και ούτω καθεξής. Επίσης, αυτές οι γυναίκες είναι εντελώς απομονωμένες, μπορεί να μένουν σε ένα διαμέρισμα μαλμια κοπέλα και η μόνη επαφή που έχουμε την πραγματικότητα με τον πραγματικό κόσμο είναι οι επαφές με τον προαγωγό, τον που είναι συνήθως ε, ο φίλος τους και έπειτα η επαφή του είναι οι πελάτε του και εμεί. Με κανέναν άλλο δεν επικοινωνούν. Και πολλέ φορέ πηγαίνουν από μια πόλη στην άλλη. Ξέρετε, μα μιλάνε, μα μιλάνε πολλέ φορέ και πολλέ φορέ μα λένε και πράγματα που δεν περίμεναν και οι ίδιε να μα πούν. Άρα τελικά μπορούμε να φτιάξουμε και τι δικέ μα αναφορέ και πιστεύω θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και το κοινωνικό σύστημα ε, στη Σουηδία, ιδίω για γυναίκε που έρχονται από μακριά ε, και πέφτουν στα ε, δίχτυα τη πορνεία. Μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Σε ό,τι αφορά την πορνεία στη Σουηδία τώρα, την ζήτηση και πώς μπορούμε να τη μειώσουμε. Φυσικά και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εξαλείψουμε την πορνεία και την εμπορία ανθρώπων στη Σουηδία. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν θα πρέπει και να εργαζόμαστε για αυτό το σκοπό με την νομοθεσία κανένα έγκλημα δεν το ε, εξαλείφουμε. Πολλά άλλα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να έχουμε εμπόδια στην αγορά σεξ. Αυτό θέλουμε να ε, πετύχουμε, γιατί αν είναι όλο και πιο δύσκολο να αγοράσει κάποιος σεξουαλικές υπηρεσίες θα σταματήσει να το κάνει. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα μπορούμε να κάνουμε. Γιατί είναι αποτρεπτικό για πολλούς άντρες αυτό. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Συμφωνώ με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Πρέπει να κυνηγήσουμε τους εκμεταλλευτές, ε, τους άνδρες που εκμεταλλεύονται ε, αυτές τις γυναίκες, ε, τις μετανάστριες. Οι κοπέλες, τα γυναίκες θα αυξηθούν, γιατί έρχονται όλο και περισσότερες μετανάστριες που είναι βάλωτες και πολύ ε, εύκολα μπορούν να πέσουν θέμα εκμετάλλευσης. Θα πρέπει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι ακόμα στο σύστημα. Και όταν ε, έρθουν σε επαφή μαζί τους ε, οι διακινητές θα τις εκμεταλλευτούν πάρα αυτά και θα βγάλουν πολλά χρήματα. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε, να το προλάβουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μωράν τώρα έχει το λόγο. Λοιπόν, εσύ. Yeah. Um, I Έχω μερικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, ανταποκρινόμενα στα σχόλιά σα, κυρία Μπίντερ, οι περισσότερε πορνίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια του τράφικινγκ όπω ορίζονται από τον ΟΗΕ. Βασικά, ο διακινητής χρησιμοποιεί εξαναγκασμό. Ε, δεν έχω δει περίπτωση πορνείας που να μην εμπεριέχει εξαναγκασμό. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα της συζήτησης προετών μεταξύ μου και άλλων γυναικών που συμμετείχαν στο εμπόριο σεξ. Ορισμένες γυναίκες λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού που δεν ανταποκρινόντουσαν αν θέλετε στον σωματέμπορο με τον ορισμό που του δίνουμε εμείς ουσιαστικά καταλάβαναν όμως την έννοια, την έννοια αυτή με συγχωρείτε ένα παιδί 15 ετών θα μπορούσε όταν ήμουν εγώ ίδια 15 ετών ε, και μπήκα στην πορνεία θα μπορούσα να επικαλυστώ ότι είμαι ε, θύμα εμπορίας σεξ διότι αυτό ανταποκρίνεται ε, στους όρους στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποίησα ποτέ και είναι θέμα πολιτιστικό τελικά το πώς κατανοεί κανείς τον κάθε όρο. Αυτό όμως που τελικά είναι η ουσία, κυρία Μπέργκερ, είναι ότι κάθε γυναίκα η οποία μπαίνει στην πορνεία ή στην εμπορία για σεξ ε, γεύεται βία. Αυτό το ξέρουμε όλες όσες έχουμε συμμετάσχει σε ένα οίκο ανοχής καθώς καθόμαστε η μία δίπλα στην άλλη, ξέρουμε ότι αυτό είναι κομμάτι της εργασίας μας τρόπον την εντός εισαγωγικών. Με τον ίδιο τρόπο ε, που άλλες γυναίκες που εργάζονται σε άλλους τομείς έχουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινέ εμπειρίες, έτσι έχουμε και εμείς αυτή της βίας. Δεν υπάρχει διάκριση λοιπόν για μένα μεταξύ πορνείας και εμπορίας είναι και τα δύο πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι που προτείνατε εσείς δηλαδή να εξεταστούν με διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας, αλλά το έχω ακούσει από αλλού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι πολύ συχνά έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι δεν θέλω να κατέβω το στραβό δρόμο και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν θέλω να δείξω έλλειψη σεβασμού, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε κάποιο βαθμό επιτρέψαμε τους εαυτούς μας και φταίω κι εγώ να πιστούμε ότι υπάρχει κάτι στραβό όταν λαμβάνει κανείς μια ηθική απόφαση. Δηλαδή η, η ηθική έγινε κάτι στραβό στη δημόσια, στο δημόσιο χώρο. Αυτό είναι γελίο όταν προέρχεται από τη γυναίκα ή τον άντρα, τον κανονικό. Μπορούμε να μπερδευτούμε όλοι πάνω σε αυτό το θέμα οι πολιτικοί μας ηγέτες τα κοινοβούλια είναι αυτά που πρέπει να διατηρήσουν, να συντηρήσουν την ακεραιότητα της σκέψης, της ηθικής και τον διαχωρισμό μεταξύ λάθους και σωστού. Ευχαριστώ. Ε, muchas gracias, eh, señora. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μωράνου. Για να ολοκληρώσουμε το πάνελ, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους όσους ήρθαν, ε, εσάς τους δύο κυρίως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς είναι η πραγματικότητα και αυτό από διάφορες σκοπιές, από διάφορες οπτικές γωνίες ε, και το αυτό το οποίο θέλουμε είναι να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό, να υπερασπίσουμε τους εμπλεκό, τις, τους, τις εμπλεκόμενες κυρίως, γιατί αφορά αυτό χιλιάδες γυναίκες. Λοιπόν, περνάμε τώρα άμεσα στην συζήτηση για το δεύτερο, στο δεύτερο πάνελ δεν έχουμε και χρόνο, γιατί ε, μέσω μιας ε, συγκεκριμένης ε, πολιτικής προσέγγισης για το φύλλο θα ακούσουμε την κυρία Μύρια Βασιλιάδου, η οποία είναι συντονίστρια του Anti-Trafficking στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να βελτιώσουμε την, ε, το συντονισμό ανάμεσα ε, στις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, του, της διεθνούς σκηνής που προσπαθούν να περιορίσουν την εμπορία των γυναικών, ελέγχει και παρακολουθεί και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την εκρίζωση της θεμοτεμπορίας, το πρόγραμμα μέχρι το 2016. Την ευχαριστούμε γιατί ήρθε εδώ και θα μας μιλήσει. Κυρία Βασιλιάδου, έχετε το λόγο. Thank you very much. Thank you Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα ξεκινώντα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει συνεργαστεί εκ του μαζί μα για τα θέματα αυτά. Όπω είπε και η κυρία Χανιμπόλ, ποτέ δεν εγκαταλείψαμε τι προσπάθειες και χρόνο με το χρόνο αποδεικνύεται αυτό και από το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Θα συνεχίσουμε. Καλωσορίζουμε την ε, πρωτοβουλία και καλωσορίζουμε και την ε, έκθεση που έχει συνταχθεί σε σχέση με την διάσταση του φίλου και θα ήθελα ιδιαίτερα για τους ε, ομιλητές και τους βουλευτές να πω ότι και η Επιτροπή έχει την ίδια προσέγγιση. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Από την αρχή υπογραμμίζουμε ότι η διακίνηση ανθρώπων σημαίνει αγορά και πώληση ανδρών, γυναικών, παιδιών, κοριτσιών, αγοριών. Από την αρχή της πρόθεσης της οδηγίας υπογραμμίζουμε ότι η σωματεμπορία είναι φαινόμενο με χαρακτηριστικά διάκρισης φύλου στηριζόμενο στην αγορά και τη ζήτηση. Και η σωματεμπορία, η λαθροδιακίνηση διαρρέει όλες αυτές, όλα αυτά τα φαινόμενα. Κοιτάξτε, δεν θα επεκτάθω σε σχέση με τους ορισμούς. Το έκανε για μένα η Κάθριν και πολύ επιτυχημένα. Την ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για λάθρεμπόριο ανθρώπων, για διακίνηση, για σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά και για πολλές άλλες ε, δυστυχώς μορφές ε, χρήσεως που έχουν να κάνουν με το φύλλο ιδιαίτερα. για εκμετάλλευση σε οικιακές βοηθούς, ε, λαθρεμπόριο παιδιών, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, λαθρεμπόριο για όργανα προς μεταμόσχευση, λαθρεμπόριο για ε, πώληση κοριτσιών ε, με το σκοπό το γάμο, ε, για υιοθεσίες. Πολλές είναι διαφορετικές μορφές. Αυτό που βλέπουμε και εντοπίζουμε από την αρχή αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον στη δική μου την ε, περίοδο υπηρεσία είναι ότι πρόκειται για μια μορφή βίαση βάρο των γυναικών. Αυτό είναι το... η σωματεμπορία. Περιορίζει τις γυναίκες και τις, γυναίκες τις και τα δικαιώματά του και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τι ευκαιρίε τη ζωή. Λέμε ότι όσον αφορά ιδιαίτερα τον περιορισμό τη ζήτηση και πρέπει να λάβουμε υπόψη την διάσταση του φύλου στο λαθρεμπόριο ανθρώπων, στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικτύου και την περιγραφή των, και τη μεταφορά στην Εθνικό Δίκαιο των Οδηγιών. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας σωματεμπορία, πρώτα απ' όλα αυξάνεται το ευάλωτο, υποδαβλίζεται η εκμετάλλευση, ε, αποτρέπεται η κοινωνική στήριξη, η βοήθεια. Όλα αυτά καταγράφονται στην έκθεσή σας. Αλλά θετικό είναι από την άλλη ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια η συζήτηση για τη διάσταση του φίλου στην ε, σωματεμπορία στην κίνηση ανθρώπων έχει λάβει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η οδηγία για το λαθρεμπόριο έχει εστίαση και στα, βήματα, και στα θύματα και στα παιδιά ιδιαίτερα και στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Και θα ήθελα να σας εξηγήσω πιο συγκεκριμένα με την ομιλία μου ότι δεν είναι μόνο λόγια αυτά που περιγράφει η νομοθεσία. Έχουμε δεδομένα στη θέση μας. Και είτε αρέσουν είτε όχι, έχουμε δεδομένα τα οποία δείχνουν τάσεις, σαφέστατες τάσεις, γιατί 80% των ε, θυμάτων που ε, διασώζονται από κάθε μορφή εκμετάλλευσης είναι γυναίκες. Ε, αυτό δεν είναι διάσταση φύλου. 95% των καταγεγραμμένων θυμάτων των υποθέσεων δηλαδή που βρήκαν, εντόπισαν ε, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι γυναίκες και 71% των θυμάτων της εκμετάλλευσης για εργασία είναι άντρες και παιδιά, αγόρια καλύτερα. Αυτό πάλι είναι διάσταση φύλου, δηλαδή το άρεν φύλο αξιοποιείται για καταναγκαστική εργασία ή σε εκμετάλλευση για εργασία. Πάλι υπάρχει διάσταση του φύλου και όλες οι άλλες συμμορφές όπου έχουμε στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες άνω του 52% στο σύνολο των θυμάτων. Θέλω όμως να προσθέσω κάτι εντός παρενθέσεως, αν μου επιτρέπετε, ότι μερικές φορές ε, φαίνεται να ε, βρίσκονται σε ανταγωνιστική θέση μεταξύ τους οργανώσεις που έχουν να κάνουν με την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων των θυμάτων. Καλό να το αποφύγουμε αυτό όλοι εσείς και εμείς να μην έχουμε ανταγωνιστική σχέση σε σχέση με την ε, εκμετάλλευση και κυρίως τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχουμε μια κινητικότητα τα τελευταία χρόνια και για τη χρηματοδότηση αλλά και για την ιδιαίτερη εστίαση στην εκμετάλλευση για λόγους εργασίας, απασχόλησης, καταναγκασμού. Γιατί αυτό τελικά μας δίνει τις απαντήσεις, την εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού ε, πρέπει να κοιτάξουμε. Βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η διακίνηση για λόγους εκμετάλλευσης ε, στην ε, σεξουαλική εκμετάλλευση συγκεκριμένα έχει καταστεί θέμα λεπτό και δεν πρέπει να συζητείτε. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού που κάποιο θύμα έχει πιο πολλά δικαιώματα από κάποιο άλλο. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δίνει τα ίδια δίκαια, δικαιώματα σε όλους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παγίως λέγει ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι παρόλες τις προσπάθειες των κρατών μελών, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ε, λαθροδιακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι έχει περιοριστεί το φαινόμενο ή είτε η σεξουαλική εκμετάλλευση είτε η διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Η διαστάση των φύλων επίσης εν προκειμένου σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε και πώς θα δίνεται η προστασία στα θύματα και πώς εξασφαλίζεται η πρόληψη από τη διάσταση του φύλου, πώς θα γίνονται οι ανακρίσεις, οι έρευνες πάλι από τη διάσταση του φύλου. Δεν θα ελπίσω στην αυτή ε, καθεαυτή συζήτηση για το θέμα της πορνείας. Ωστόσο λέγεται ότι είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και δεν μπορεί κανείς να λέει ότι είναι παράγον υψηλού κινδύνου για το, η λαθροδιακίνηση ή η πορνεία. Εγώ δεν βλέπω τίποτε το λεπτό ή ευαίσθητο εδώ πέρα. Εφόσον οι αστυνομικέ αρχές μου λένε ότι τα θύματα, σχεδόν όλα τα θύματα της ε, λάθρο διακίνησης ανθρώπων σωματιμπορίας καταλήγουν στην πορνεία, τότε θεωρώ ότι είναι ζήτημα υψηλής διακινδύνευσης. Είναι τομέας υψηλής διακινδύνευσης όπως είναι και η αλία για, το, για τον αλία. Δεν θα μου πει κανείς ότι ε, ακούμπησε κάποιο ταμπού εάν ισχυριστώ κάτι τέτοιο, όπως και για τη λαθροδιακίνηση. Είναι η λαθροδιακίνηση υψηλού επίπεδου υψηλής σηματοδότησης κίνδυνο για την πορνεία. Ποσοστά. Τι σημαίνουν τα ποσοστά. Πιο πολλά εδώ, πιο πολλά εκεί. 16% από τα καταγεγραμμένα, σημειώνω καταγεγραμμένα πάντα θύματα, μας λέει η Eurostat, είναι παιδιά. Τι θα πούμε λοιπόν. Μόνο 16%. Ε, καλά εντάξει, δεν πειράζει. Δηλαδή μόνο νούμερα κοιτάμε. Δεδομένα. Ή κοιτάμε τον άνθρωπο. Μίλησαν οι συνάδελφοι ε, για την διακίνηση για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλούμε και για άλλο τύπου εγκλήματα, πολλαπλούς βιασμούς. Μπορεί να γίνεται λόγος για το βιασμό όταν κάποιος υποχρεούται σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς να έχει δώσει τη συνένεσή του. Αλλά όταν μιλάμε για θύματα, και μην με παρεξηγήσετε, Νομίζω ότι όταν φτάσει η ώρα να μιλήσουμε για τα θύματα είναι αργά πια. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το θύμα ήδη έχει φερειπίνει σεξουαλική εκμετάλλευση, ε, πέσει θύμα βιασμού. Ίσως και χιλιάδες φορές. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι οι ίδιοι έχοντας συνομιλήσει με τα θύματα και τα παιδιά ακόμα που έχουν πέσει θύματα ε, αγοραπολωσίας που έχω δει εγώ και έχω ρωτήσει ένα κορίτσι, το ανέφερα και τις προάλλες, 15 ετών, τώρα με κόρη δύο ετών που προέκυψε στεραποβιασμό και τη ρώτησε τι θα κάνω. Τη ρώτησα τι θα κάνεις στο υπόλοιπο τη ζωή σου, τι θες να κάνεις και η ερώτηση με την οποία μου απάντησε ήταν ποια ζωή. Και θα συμφωνήσω μαζί σας εδώ ότι η δουλειά μας είναι να προλαμβάνουμε. Η πρόληψη είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για να μην φτάνουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία με μεγάλη καθυστέρηση. Και σημειώνω αυτό που είπε η Ρέιτσελ για τον τελικό στόχο της ε, σωματεμπορίας που είναι η πορνεία. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι τα θύματα έχουν δικαιώματα. Είναι δικαιούχοι. Υποκείμενα δικαιωμάτων. Και με ενοχλεί πολύ ο όρος και με εξοργίζει ο όρος του trafficked person, ότι δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος έχει μπει λαθρέα και δεν έχει κανένα δικαίωμα. Όχι, είναι ένα θύμα λαθρέας διακίνησης και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να προσφέρουμε την εσφάλιση των δικαιωμάτων τους. Έχουμε την νομοθεσία για την καταπολέμηση της διακίνησης, ε, τη στρατηγική της σχετική, σας τα έχω ήδη παρουσιάσει, από τις λεπτομέρειες. Είναι σαφές όμως ότι η διάσταση του φύλου είναι πολύ έντονη και στα δύο αυτά εργαλεία. Τι σημαίνει όμως λαθροδιακίνηση. Η κυρία Μπέρντερ σαφώς περιέγραψε το νομικό ορισμό. Για μένα όμως η λαθροδιακίνηση αυτή είναι μια απλή έννοια. Για μένα είναι το να κερδίζει κανείς χρήματα σε νόμιμο ή και παράνομο τομέα και να υπάρχει η ζήτηση. Εάν δεν υπάρχει ζήτηση, αν κανείς δηλαδή δεν έρχεται να στήσει να υπάρχει αυτό θύμα της εκμετάλλευσης, ή αν δεν υπάρχει το κέρδος, αν βγει η ζήτηση και το κέρδος, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες φρικτές και αποτρόπες καταστάσεις ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να είναι λαθροδιακίνηση. Άρα πρέπει να κοιτάμε πού πάει το χρήμα, πρέπει να ψάχνουμε ποιος και σε ποιο επίπεδο και σε ποιο είδος της διαδικασίας ε, οδηγεί στο να χάνεται το ίχνος του χρήματος. Η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας μας λέει ότι μπορεί να έχει φτάσει και τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε νόμιμους χώρους εργασίας ή καταναγκαστική εργασία. Για να δούμε και τους παράνομους η ζήτηση επίση, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση νομικά να περιορίσουν και να αποθαρρύνουν τη ζήτηση και να ενισχύσουν τη συνειδητοποίηση του φαινομένου. Η δουλειά μου είναι να επιβλέπω την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου και πρέπει να το επαναλαμβάνω αυτό συνέχεια. Τα κράτη-μέλη μα ζητούν ε, να εξετάσουμε το ζήτημα τη ποινικοποίηση εκείνων που αξιοποιούν το δίκτυο τη λαθροδιακίνησης γνωρίζοντα ότι το αντικείμενο τη ολική είναι θύμα. Το κάνουμε και θα επανέλθω σε αυτό. Στη στρατηγική. Διαρκώς καλούμε να παρακολουθείτε το ίχνος του χρήματος. Και αν μπορέσω να εκθέσω περισσότερο τις θέσεις μου, το χρήμα είναι αυτό το οποίο καθοδηγεί τη ζήτηση και η ζήτηση αντίστοιχα καθοδηγεί το χρήμα. Νομίζω ότι μπορεί να δοθεί και μια καλύτερη εξήγηση αργότερα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει πως και στην, στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση και στο θεματολόγιο για την ασφάλεια εξετάζεται η λαθροδιακίνηση των ανθρώπων γιατί εκεί στην ασφάλεια ιδιαίτερα είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει το χρήμα, υπάρχει η εκμετάλλευση των ανθρώπων και το φαινόμενο της διάχυσης από το οργανωμένο έγκλημα και σε άλλους τομείς. Και θα πω, μια και το έθιξαν οι ευρωβουλευτές ε, για, για τη λαθροδιακίνηση, Έχουμε στοιχεία από τη συλλογή πληροφοριών, από τις υπηρεσίες των πληροφοριών. Ξέρουμε ότι τα πλοία αυτά που φέρνουν τους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους ε, που φεύγουν πρόσφυγες για να έρθουν στην Ευρώπη μεταφέρουν και νεαρά κορίτσια από την Αλγερία. Άρα η λαθροδιακίνηση μπορεί να ισοδυναμεί με σωματεμπορία. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι οδοί της, ε, λαθρεμπορία, της λαθροδιακίνησης αξιοποιούνται από τις ε, σωματεμπόρους και τα δίκτυά τους, όπως στην περίπτωση της νοικηρίας. Και ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω εδώ το ενδιαφέρον που έχει δείξει στο σώμα ε, για την προστασία των παιδιών που έχουν θύματα αυτών των δικτύων και κάθε μορφής εκμετάλλευσης κυρίως σεξουαλικής. Ξέρουμε ότι ξεκινάνε παιδιά και μένουν θύματα και σε όλη την ενήλικη τους ζωή. Η αφελής μου όμως ερώτησης θα είναι το εξής. Άδικο, άδικο που με περιορίζετε. Ε, εάν έρθει, αν μεταφέρει κάποιος ένα παιδί στην Ευρώπη, 4 με 8 χιλιάδες ευρώ είναι η αξία ενός παιδιού που θα μεταφερθεί στην Ευρώπη. Μπορεί να φτάσει και 40.000 ευρώ η αξία, η αγοραία αξία ενός παιδιού. και αμφιβάλλω κάπως για το εάν αυτό το τίμημα αντιστοιχεί μόνο σε εξαναγκασμό στην επαιτία στους δρόμους τα πρωινά. Έχω μόνο δύο λεπτά στη θέση μου, δεν μπορώ να επεκταθώ. Αλλά έχω μια μελέτη που δημοσιεύεται αφορά τις ομάδες υψηλού κινδύνου, κυρίως τα παιδιά, ως θύματα και σεξουαλικής εκμετάλλευσης που συνεχίζεται και όταν ενηλικιώνονται, πόσα υπάρχουν τα, τα μοτίβα της βίας της βάρος γυναικών και παιδιών, η ε, διακριτική μεταχείριση των φύλων, ε, θυματοποίηση κτλ. Έχουμε δημοσιεύσει την έκθεση αυτή, είναι διαθέσιμη στο δικτύο μας τα και δύο εβδομάδες και το πρώτο πρέπει να κοιτάξει κανείς είναι η έκθεση τάσεων δύναμη του άρθρου 20 τα κράτη-μέλη μου αποστερούν τις εκθέσεις τους για τις εξελίξεις σχετικά με το σωματεμπόριο και ε, διατυπώνουμε τώρα την έκθεσή μας που είναι έτοιμη για το Μάρτιο του 2016 επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης την έκθεση με το άρθρο, δυνάμει του άρθρου 23 για την μεταφορά σε εθνικό του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Θέλουμε να ακούσουμε αντίστοιχα και τις θέσεις του Κοινοβουλίου και για να ολοκληρώσω η οδηγία κατά του ισοματοπορίας έχει ε, από την κοινοποίηση που μας έχει γίνει μετατεθεί σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό δίκτυο πλην της Γερμανίας. Αυτή δεν μας έχει κοινοποίησει μεταφορά στο εθνικό δίκτυο. Επίσης, στον τελικό χρήστη, στην πρόληψη, στην παρακολούθηση του, της υπόθεσης ε, με κατάλληλες ε, προτάσεις συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έχουμε μια οδηγία για τις κυρώσεις όπου ε, ποινικοποιείται η εν γνώση του χρήστη αξιοποίηση σεξουαλικών υπηρεσιών υπηκών τρίτων κρατών. Πρέπει να διευρυνθεί το έργο αυτό και προσπαθώντας να κλείσω κυρίες και κύριοι, είναι πολλές περιπτώσεις όπου δεν ε, απαγορεύεται η αγοραπολισία ανθρώπων και η αξιοποίηση των υπηρεσιών των ανθρώπων που, πέσουν θύματα, που πέφτουν θύματα αγοραπολισίας. Μπορεί να το κάνουμε δηλαδή και να μην μας τιμωρήσει κανείς και έχω ρωτήσει 500 φορές. Μέχρι κάποιο να μου απαντήσει θα το ξαναρωτάω. Έχω ρωτήσει εισαγγελείς, ε, ανακριτές, δεν έχω πάρει απαντήσεις. Ξέρετε να υπάρχει άλλο τομέα εγκληματική δραστηριότητα όπου ο αξιοποιών την εκμετάλλευση δεν μπορεί να προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Και αν υπάρχει αυτό, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή λέμε ότι μπορεί κανείς να αγοράζει και να πολλοί ανθρώπους και να αξιοποιεί τις υπηρεσίες, να εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες αυτών που αγοράζονται και πουλούνται. Αυτό είναι το μήνυμα στην κοινωνία. Ο νόμος έχει ρυθμιστικό αποτέλεσμα και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Χρειαζόμαστε τον νόμο για το θέμα του περιορισμού της ε, ζήτησης είχαμε την ε, ημέρα για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας και ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές που ήρθαν. Κάποιοι μας ρωτούσαν γιατί μιλάτε για περιορισμό της ε, ζήτησης, είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Α, όχι, με συγχωρείτε, είναι το άρθρο 18 της οδηγίας. Και γιατί καλέσατε, λέει, αυτούς τους ανθρώπους, κάλεσα αυτούς που δουλεύουν πάνω στο αίτημα της, του περιορισμού της ζητήσεως και για να τιμήσουμε το πνεύμα της οδηγίας και της γενικές κατευθύνσεις, η Επιτροπή πρώτη ξεκίνησε μία μελέτη για να αντιληφθούμε καλύτερα το φαινόμενο με το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ που ανέλαβε την μελέτη και έχουμε και εκπρόσωπο σήμερα εδώ και εδώ επανέρχομαι στα σχόλια της κυρίας Χόνιμπολ για το ψήφισμα του 2014 πάνω στο, γύρω από το οποίο περιστράφει η μελέτη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να σας κάνουμε παρουσίαση. Βέβαια η Σίλβια από το Πανεπιστήμιο του Λάγκαστερ να σας πει περισσότερα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, για 10 ακόμα δευτερόλεπτα θα σας κρατήσω. Δεν υπάρχει θέμα που να είναι λιγότερο σημαντικό από τα άλλα. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε ποιο θέμα είναι σημαντικό ή ποια μορφή εκμετάλλευση έχει μεγαλύτερη σημασία από τι δεν ε, είμαστε σε ανταγωνιστική σχέση, σχέση με τις μορφές εκμετάλλευσης και δεν υπάρχει ευαίσθητη μορφή εκμετάλλευση. Δεν είναι ευαίσθητο θέμα η συζήτηση της κατάφορης εκμετάλλευσης και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά υπάρχει ανάγκη για κατεπίγουσα δράση. Πολλέ φορέ κάποιο μπορεί να ξεκινήσει θεωρώντα ότι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του, αλλά δεν τα καταφέρνει ποτέ, σα διαβεβαιώ, και πρέπει να θυμόμαστε πάντα αυτό το γεγονό και τα δικαιώματα των θυμάτων. Έχουμε ευθύνη να αποδώσουμε δικαιοσύνη στα θύματα. Και αν δεν ρωτήσουμε ποιο κερδίζει, ποιο αξιοποιεί τι υπηρεσίε, καλύτερα να κλείσουμε το μαγαζί και να γυρίσουμε σπίτια μα, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Muchas gracias, señora Ευχαριστώ πολύ κυρία Βασιλιάδη και λυπάμαι πολύ που περιορίζω το λόγο και κλείνω το μικρόφωνο τελικά σχεδόν ε, στους ομιλητές. Απλά θέλω να δώσω το λόγο σε όλους όσους ε, έχουν έρθει εδώ και γι' αυτό θα περάσω ευθύ αμέσω στην κυρία Σίλβη Γουόλμπι, καθηγήτρια κοινωνιολογίας που είναι και στην ε, UNESCO, πρόεδρος ε, της έρευνας φίλου, στο Πανεπιστήμιο του Λάγκαστερ εργάζεται, έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που άπτονται της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Αντιτράφικινγκ. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα να σας ε, ε, ξαναδούμε σε σχέση με το έργο το οποίο επιτελείται. Σας δίνω αμέσως το λόγο κυρία Βόρντι. Thank σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα που είμαι εδώ για να συμβάλλω όσον αφορά το έργο των πανεπιστημίων στην δημοκρατική, στον δημοκρατικό διάλογο, στη δημοκρατική ακρόαση. Θα σας αναφέρω θέματα τα οποία αφορούν το θέμα του φύλου στο τράφικινγκ. Θα κάνω δύο πράγματα. Θα σας προσφέρω νέους τρόπους σκέψης σε σχέση με τη διάσταση του φύλου στο τράφικινγκ. Ακόμη θα σας προσφέρω κάποιες συστάσεις συμπληρωματικές. Ε, η έκθεση για την οποία, στην οποία αναφέρομαι, όπως είπε η Μέρη, θα δημοσιευθεί. Αφορά το τράφικινγκ ανθρώπων. Έχουμε μια πανευρωπαϊκή ομάδα που εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Έχω τρεις συναδέλφους που είναι εδώ από άλλα πανεπιστήμια ε, που συνεργάζονται ακριβώς στη σύνταξη αυτής της έκθεσης από τη Γερμανία κτλ. Ασχολούμαστε βασικά με το θέμα της πρόληψης καθώς και με το θέμα της διάστασης του φύλου. Η πρόληψη είναι στην καρδιά της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην καρδιά της σχετικής οδηγίας. Τώρα, πώς αντιλαμβανόμαστε την πρόληψη. Θα σας προτείνω να ξεχάσετε τη σκέψη σας ότι η πρόληψη αναφέρεται στις επιλογές των ατόμων. Ε, σκεφτείτε μάλλον τα θέματα όσον αφορά τις ρυθμίσεις που επιβάλλονται από τους θεσμούς, ειδικότερα από τους κερδοσκοπικούς θεσμούς. Λοιπόν, ας περάσουμε από το άτομο στους θεσμούς. Ε, οι θεσμοί είναι αυτοί που ρυθμίζουν και εσείς ρυθμίζετε τους θεσμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αντιλαμβάνεται την ισότητα των φύλων. Είναι διακριτή διακριτός αυτός ο τρόπος, είναι εμπεδωμένος και συνεχίζει. Μιλάμε δηλαδή για ίση μεταχείριση όταν μιλάμε για την ισότητα των φύλων και αυτό συνεπάγεται εξειδίκευση του φύλου. Εάν δεν υπάρχει εξειδίκευση του φύλου δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίση μεταχείριση. Ακόμη έχουμε αρχές ισορροπίας των φύλων, στη λήψη των αποφάσεων, ενσωμάτωσης των φύλων στους μηχανισμούς και αυτές οι αρχές ισότητας των φύλων εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πολιτικών ώστε να υπάρχει συνέπεια και συντονισμός της πολιτικής για την κατάργηση του τράφικινγκ. Λοιπόν, θα μιλήσω για κάθε παράμετρο. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για την υποστήριξη των θυμάτων. Καμιά φορά αυτό αντιμετωπίζεται σαν να είναι το τελικό πράγμα που πράττουμε όταν βοηθούμε ένα θύμα. Αλλά ουσιαστικά η βοήθεια προς το θύμα, αν είναι σωστή, μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή και στην πρόληψη. Δηλαδή, με πολύ απλό τρόπο ε, προλαμβάνεται την επανάληψη των θυμάτων υποστηρίζοντας καλά τα θύματα διότι τα θύματα αυτά που τα υποστηρίξατε σωστά μπορούν να εκφραστούν στον δημόσιο διάλογο βάσει των εμπειριών τους. Το βάθος της βοήθειας που δίνουμε στα θύματα είναι πραγματικά σημαντικό. Έχουμε διάφορες λεπτομερείς συστάσεις στην έκθεσή μας. Δεν θα σας την διαβάσω αυτή τη στιγμή, αλλά αφορούν αυτό το θέμα. Τώρα, η δίωξη. Η δίωξη. Η δίωξη λοιπόν δεν είναι αυτός ο σκοπός, αν και οπωσδήποτε είναι σημαντικό μέσα στο μηχανισμό της δικαιοσύνης. Μειώνοντας την ατιμορρησία μπορείτε να οδηγήσετε σε πρόληψη. Αυτό είναι το ζήτημα. Καμιά φορά η δίωξη αντιμετωπίζεται ε, μόνο σε θέματα ποινικά. Εμείς συστήνουμε να περιλάβετε όλο το φάσμα των ενιών δικαίου και να μην περιοριστείτε μόνο στο ποινικό δίκαιο. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν ε, πρακτικές νομικές που έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν ε, καταδειχθεί αποτελεσματικές. Το ποινικό δίκαιο αναμφίβολα είναι ο ακρογωνιαίος λήθος, η βάση του δικαίου. Αλλά δεν είναι το μόνο δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε και σε αυτό το θέμα συγκεκριμένες συστάσεις, διατυπώσεις. Τώρα, θα ήθελα περισσότερο να επικεντρωθώ στον πιο παραδοσιακό τομέα πρόληψης που αφορά τη ζήτηση. Να αποθαρρύνει κανείς και να μειώσει τη ζήτηση που οδηγεί σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρόκειται, Πρόκειται για το άρθρο 18 της οδηγίας. Λοιπόν, πρέπει να ξανασκεφτούμε τη ζήτηση. Πολύ συχνά περιοριζόμαστε στη σχέση μεταξύ των ατόμων πολιτών και των ατόμων αγοραστών. Αλλά παραγνωρίζουμε το πιο σημαντικό μέρος που είναι οι θεσμοί που επικεντρώνονται στην κερδοφορία. Λοιπόν, υπάρχει μία ολόκληρη σειρά από τρίτα μέρη, πολύ σημαντικά, τα οποία κάπου εξαφανίζονται επειδή έχουμε ε, επειδή η συζήτηση έχει πολλωθεί και συνεπώς εμείς προτείνουμε να επανέλθουμε στο θέμα της ρύθμισης των κερδοφόρων θεσμών και αυτό το θέμα να το βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης και όχι να το παραμερίσουμε. Τα τρίτα μέρη δηλαδή που επωφελούνται από όλα αυτά. Υπάρχουν πολλές εμπειρίες στην Ευρώπη ως προς την πρόληψη και την ρύθμιση κλάδων που έχουν σχέση με το, με το Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ποικιλομορφία από τη Σουηδία, Γερμανία κτλ. και τις καινοτομίες. Για μας τους ακαδημαϊκούς πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φυσικό πείραμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Πρέπει να χαιρόμαστε για την καινοτομία στην Ευρώπη. Αυτό το τρίγωνο από τη συνάδελφο και φίλ Colin Σάουερ μας δείχνει πώς σκεφτόμαστε για τη ρύθμιση της πορνείας σε σχέση σε σχέση με τους υπόλοιπους φορείς. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μόνο η σχέση μεταξύ του ατόμου αγοραστή και του ατόμου πολιτή, αλλά έχουμε τη σημαντική έννοια αυτών που αποκομίζουν τα κέρδη, κέρδη τώρα, μέσω μισθωμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, παραδείγματο χάρη, αλλά παρόλα αυτά αυτό σημαίνει κέρδη που αποκομίζουν από, αυτό από αυτή τη σχέση. Υπάρχουν, ε, υποτιμούνται όλα αυτά πρέπει να πω. Και έχω δύο λόγια να πω σε σχέση με μια εμπειρία στη Γερμανία και τις κάτω χώρες που έχει παρανοηθεί. Καμιά φορά περιγράφεται σαν απλή αποποινικοποίηση. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντική αύξηση της ρύθμισης του χώρου του Έχουμε δει μερική από ποινικοποίηση και αύξηση της ρύθμισης ταυτόχρονα. Η δημοκρατική συζήτηση σε αυτά τα κράτη-μέλη έχουν συζητήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις καινοτομίε. Έχουμε δει ήδη εξελίξεις που προσημιάζουν με εξελίξεις και στη Σουηδία. Θα πρέπει λοιπόν να ρίξετε μια ματιά σε αυτές τις λεπτομέρειες για να αποφύγουμε την υπερεκμετάλλευση που υπάρχει σε ορισμένες, ορισμένους τύπους ε, πορνείας. Ένας τρόπος είναι η πλήρης απαγόρευση. Απαγορεύεται η πορνεία στον δρόμο. Ε, ε, χρησιμοποιούν μεγάλους μηχανισμούς για να το εφαρμόσουν και σε συγκεκριμένες πόλεις. Ταυτόχρονα λένε ότι οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτε, ευάλωτοι και έστω και αν ενηλικιώνονται στα 18, αυτό είναι πολύ νωρίς για την πορνεία. Και συνεπώς μπορεί κανείς νόμιμα να αγοράσει σεξ όχι στα 18 αλλά στα 21. Έχουμε λοιπόν μία ρύθμιση η οποία προκύπτει προκύπτει κάτω από δημοκρατική πίεση που επιβάλλει τύπους και μορφές πορνείας σε χώρες που καμιά φορά εμφανίζονται σαν να είναι χώρες απελευθέρωσης από τις ρυθμίσεις. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι νομίζετε. Αυτό το οποίο λέμε εδώ είναι ότι η ζήτηση δεν αφορά μόνο τους άμεσους καταναλωτές, αφορά και όλους όσους εποφελούνται από την ιστορία αυτή, γιατί το τρίγωνο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Όπως είπε και η Μύρια, Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ποινικοποίηση της αγοράς, πώς θα δούμε την, πώς διαμορφώνεται η σχέση με την Σουηδία. Δεν θα έχω χρόνο να πω σε λεπτομέρειες, αλλά είδατε τι γίνεται στη Σουηδία. Αυτό το οποίο πρέπει να ξανασυζητήσουμε είναι η ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ συχνά οι συζητήσεις μας έλκονται, αν θέλετε, από το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Όμως προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική. Εμείς στην Ευρώπη συστηματικά έχουμε αποποινικοποιήσει την πώληση του σεξ. Έχουμε αποποινικοποιήσει την αγορά και έχουμε υποτιμήσει τις αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα σε όλες τις ευρωπαϊκές ενώσεις και έχουμε διαφοροποιήσει την αποπενικοποίηση της ε, ε, πώληση ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν διατηρήσει την ποινικοποίηση της ε, κερδοφορίας αν θέλετε από τις υπηρεσίες ΕΞ. Οι περισσότερες χώρες θεωρούν ότι είναι παράνομο να ε, εκμεταλλεύονται τους πόρους που προέρχονται από την πορνεία άλλων. Επομένως, τι εννοούμε όταν λέμε εκμετάλλευση της πορνείας, των, των καρτών της πορνείας, όταν μιλάμε για μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Πρέπει να, λάβουμε, να βαίνουμε υπόψη μας και αυτούς οι οποίοι πολλούν αυτές τις υπηρεσίες. Στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ποινικοποιείται και η εκμετάλλευση των άλλων και, ε, ε, και το κέρδος που αποκομίζεις από την εκμετάλλευση των άλλων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι λέει η οδηγία και, τα, και το πρωτόκολλο. Ε, οι Αμερικανοί δεν έχουν αυτού του είδους ε, νομοθετικές διατάξεις. Επομένως αυτό το οποίο λέει και η Διεθνής Αμνηστία μιλά, μπερδεύει λίγο την ε, αγορά και πώληση υπηρεσιών του σεξ με την εκμετάλλευση και την, και την την ίσπραξη, αν θέλετε, κέρδους από αυτές τις ε, υπηρεσίες. Έχουμε βάλει δηλαδή εμείς ένα, μια απόχρωση, αν θέλετε, στις ε, νομοθετικές μας ε, διατάξεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις. Η, πόλη, η πρόληψη τώρα και η, η συνοχή της πολιτικής. Πολλές φορές Αυτά τα δύο αντιμετωπίζονται σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Όμως, εάν εφαρμοστούν ε, συστηματικά σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη σωματεμπορία, αλλά στην ασφάλεια, εξωτερικές σχέσεις ε, και εσωτερική αγορά, τότε θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να γενικεύσουμε τις συνέπειες ε, των δεσμεύσεών μας όσον αφορά τις φιλετικές διακρίσεις και έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλουμε να πούμε για το πώς ε, θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε και να αλλάξουμε τις δομές ε, της, για, την, ε, για τις διαφορές των φύλων που δεν στηρίζονται σε εκμετάλλευση, σε, στο κέρδος, ε, και στην ε, ε, εκμετάλλευση λόγω σωματεμπορίας άλλων. Έχουμε συγκεκριμένους τομείς για τους οποίους κάνουμε συστάσεις, ζητάμε να γίνουν μετρήσεις γιατί χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα, χρειαζόμαστε μια συνοχή όλων αυτών των αρχών που διέπουν τις πολιτικές μας και τα προγράμματα, προγράμματα δράσης μας. Ε, πιστεύω ότι αν λάβουμε υπόψη μας τις διακρίσεις των φίλων σε όλους τους τομείς, τα πράγματα ε, θα προχωρήσουν καλύτερα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία ήταν πολύ θετική αποποινικοποιήσαμε την πώληση αλλά δεν αποποινικοποιήσαμε την εκμετάλλευση τρίτων. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και ποιος είναι ο γενικός μας στόχος, ότι θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την σωματεμπορία και την παράνομη διακίνηση των ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλές ε, προτάσεις ε, έχουμε, ακούσαμε, έχουμε μία, μέχρι τις μία και πέντε τους διερμηνείς. Ε, αν θέλουμε να συνεχίσουμε μετά, θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Η κυρία Μπεκαρίλα ζήτησε το λόγο όμως. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω της εισηγήτριες και να ζητήσω ε, από την ε, συντονίστρια του anti-trafficking ε, που την γνώριζω πολύ καλά, την κυρία Βασιλιάδου. Και για να ενημερώσω ενδεχομένω και τους υπόλοιπους. Δεν θέλω να σας πω ότι όταν ασχολήθηκα αυτά τα έξι χρόνια ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο είδα ότι πολύ λίγα είναι γνωστά για τα θύματα και μιλάω γενικά όχι απλά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή οποιοδήποτε ε, θύμα. Το δικό μου υπόβαθρο είναι διαφορετικό. Ε, ασχολήθηκα πιο πολύ με τα θύματα τρομοκρατίας, ε, αλλά πάντοτε με ενδιαφέρει και πάντοτε ασχολούμαι με τα υπηρεσίες παροχής, υποστήριξη στα θύματα κτλ. Και επειδή λοιπόν εργάζομαι σε σχέση με τα θύματα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει το European Protection Order, εγκρίθηκε το σχετικό νομοθέτημα και έπειτα είχαμε και την οδηγία για την υποστήριξη, την προστασία και τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόπινων πράξεων. Το European Protection Order, αυτό το ένταλμα προστασίας, είναι αν κάποιος ε, για κάποιον ε, εντολή, ασφαλιστικά μέτρα και δεν μπορεί να πλησιάσει, παραδείγματο χάρη, ε, κάποιο άλλο άτομο, να ισχύει και για το θύμα να υπάρχει προστασία και στις άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες, διότι ε, μέχρι τώρα έπρεπε να αρχίσει ένα θύμα από το μηδέν, να πρέπει να αποδείξει, να φέρει στοιχεία για να μπορεί να προστατευτεί. Αν λοιπόν ε, μια γυναίκα που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλης εκμετάλλευσης έπρεπε να περάσει από δικασία, Πολλές φορές τη δολοφονούσε ο, η ε, θήτης και μετά, επομένως δεν είχε κανένα νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Και έχουμε και μια άλλη οδηγία η οποία υλοποιείται αυτή τη στιγμή, έχουν πέρασει τρία χρόνια που ήταν μεταβατική περίοδος ε, και πλέον πρέπει να τεθεί σε ισχύ. Και το ερώτημά μου είναι, η συντονίστρια κατά της εμπορίας, τι θα κάνει γιατί υπάρχει σε αυτή την οδηγία ε, δεσμέτρων, αναφέρονται τα θύματα σωματεμπορίας, ε, οι γυναίκες συγκεκριμένα, τα θύματα σωματεμπορίας. Και θα ήθελα και αναφέρομαι και στον κύριο Χέντριξεν εδώ, η αστυνομία. Γνωρίζει κάτι για αυτή την οδηγία που γίνεται λόγος αυτήν για κατάρτιση, εκπαίδευση της αστυνομίας, εκπαίδευση των δικαστικών και επειδή μιλάμε για θύματα σε μια άλλη χώρα. Τι γίνεται όταν κάποιος καταγγέλει ε, μια εξωτερική πράξη χώρα, ε, σε μια άλλη χώρα και στη χώρα καταγωγής τους. γιατί δεν θέλουμε να υποστεί δεύτερη θυματοποίηση το θύμα και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Βασιλιάδου που είπε ότι όλα τα θύματα είναι τα ίδια, έχουν την ίδια ε, σπουδαιότητα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε συγκεκριμένα αν έχετε κάποιοι κάτι να μας πείτε και θα ήθελα επίσης να μου πείτε και τι γίνεται με τις γυναίκες και τα παιδιά στους καταβλισμούς προσφύγων και γενικότερα με αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα που έχουμε υπάρχουν και βιασμοί και κακοποίηση και αγοραπολισίες παιδιών θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες αν έχετε. Και τέλος να πω στην κυρία Μωράν ότι ε, δεν θα μπορούσα να δώσω περισσότερο ε, με τα λόγια με τα οποία κλείσατε την δευτερολογία σας. Δηλαδή ότι το ουσιώδες είναι να καταλάβουν και να καταλάβουν και οι πολιτικοί ε, τι θα πει καλό και τι θα πει κακό. Νομίζω ότι αν κάναμε αυτή τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα και το βλέπουμε αυτό στον κόσμο των θυμάτων. Είμαι και εγώ θύμα, θύμα τρομοκρατίας και πραγματικά όταν μιλάτε, μιλάτε κατευθείαν στην καρδιά μου. Δεν ξέρω αν οι άλλοι ε, μπορεί να το καταλάβουν τόσο όσο εγώ που έχω υπάρξει θύμα. Κάποιες φορές ε, το βλέπω. Δεν ξέρω τι φταίει, μπορεί να φταίει το παρελθόν μου. Εγώ πάντως είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τα θύματα τα δικαιώματα των θυμάτων, αλλά πράγματι όταν ακούω τέτοια λόγια ε, με αγγίζουν. Και οι γυναίκε, ξέρετε, δεν έχουν ούτε χρήματα ούτε δυνατότητα άσκηση πίεση. Λίγη δύναμη έχουν στη δεσή του. Ε. Και αυτό ίσω είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε του διερμηνεί. Θα σταματήσει εδώ η διερμηνία και θα δοθούν οι απαντήσει από εδώ και πέρα στα αγγλικά